Uh, um, Καλημέρα σας. Ε, βλέπω ε, λίγους σήμερα το πρωί εδώ. Θα ήθελα να σας ε, καλωσορίσω και χαίρομαι που είναι εδώ και ο εισηγητής μας για το πρώτο θέμα και ελπίζω λίγο περισσότεροι θα εγκαταλείψουν τη διακάδα έξω για να έρθουν εδώ στη συζήτηση. Πάντως θέλω να σας καλωσορίσω και θέλω να καλωσορίσω και όσους μας ακούν από το διαδίκτυο. Καλώς ορίσατε στη συνεδρίασή μας ένα υπέροχο για όλους το πρωινό ε, στις Βρυξέλλες όμως ε, δυστυχώς εμείς εδώ δεν έχουμε παράθυρα στην αίθουσα και μάλλον γι' αυτό τόσο πολύ λείπουν. Έχουμε βέβαια φορτωμένη ημερησία διάταξη τις επόμενες ε, δύο ημέρες της συνεδρίασης και έχουμε και τη σημαντική αναθεώρηση της έκθεσης του κυρίου Τεραμπέλα για τις δημόσιες συμβάσεις σήμερα το απόγευμα και είναι ένα από τα μεγάλα θέματα επί των οποίων εργαζόμαστε, αλλά έχουμε και άλλες σημαντικές γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις ε, νομοθεσίας και μη νομοθετικές εκθέσεις να εξετάσουμε. Λοιπόν, να κάνω κάποιες ανακοινώσεις ε, σχετικά με τις διαδικασίες. Ε, καταρχήν, να εγκρίνουμε επίσημα την ημερήσια διάταξη θα γνωρίζετε ότι την έκθεση της κυρίας Μακλάρκιν την αλλάξαμε σήμερα με της κυρίας Χάνσες που, είναι, που αφορά το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η έκθεση της κυρίας Χάνσες για την ε, επιχειρηματική πρωτοβουλία θα συζητηθεί αύριο. Και μια σημαντική ανακοίνωση είναι η εξή. Να σας γνωστοποιήσω ότι δεν θα υπάρξει ψηφοφορία όπως έχει προβλεφθεί για την πιθανή εντολή ε, διαπραγματεύσεων ε, με το Συμβούλιο για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία, αλλά θα έχουμε μία έκθεση για ένα ψήφισμα από τη Μαζί Επιτροπή για το Single Market Act και τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη. Και αυτό ε, από κοινού μαζί με μια σχεδιαζόμενη δήλωση από τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, τον κύριο Μισελ Μπαρνιέ, την Τετάρτη, 13 Ιουνίου στο Στρασβούργο, πιθανότητα το απόγευμα ή μάλλον ε, σίγουρα το απόγευμα θα ε, μας παρουσιάσει δύο σημαντικές εκθέσεις για την εφαρμογή της οδηγίας για τις επιχειρήσεις, τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση της εσωτερικής αγοράς, της ενέας αγοράς και ιδέες για το επόμενο στάδιο για το Single Market Act και το ψήφισμα μας ε, θέλει να παρουσιάσει κάποιες ιδέες που θα συμπεριληφθούν για το πρόγραμμα 2013 πριν η Κομισιόν ολοκληρώσει το έργο της ε, για το θέμα αυτό. Δεν είχαμε χρόνο για πληρή έκθεση, έτσι λοιπόν επιλέξαμε αυτή την οδό. Τώρα, σε σχέση με το ψήφισμα που ε, με το οποίο ασχολήθηκαν όλε οι πολιτικέ ομάδε. Έκαναν πολλή δουλειά και σα ευχαριστώ και μα υποστήριξε και η σκληρά εργαζόμενη γραμματεία. Το σχέδιο κειμένου λοιπόν αυτού θα είναι διαθέσιμο σήμερα το πρωί αργότερα. Θα το μοιράσουμε σε όλου, έτσι όλοι θα έχετε τη δυνατότητα να το εξετάσετε πριν από την ψηφοφορία. Λοιπόν, αυτό ήταν σημαντική πληροφορία για κάποια άλλα θέματα τώρα στου φακέλου σα. Έχετε την ετήσια έκθεση του 2011 για το σύστημα ειδοποίησης ε, για τα επικίνδυνα προϊόντα. Ε, το παρακολουθεί αυτό το θέμα πολύ, από πολύ κοντά η Επιτροπή και ε, έχουμε και την εισηγήτρια για την γενική ασφάλεια ε, των ε, προϊόντων. Ε, θα έχουμε αναθεώρηση στο φθινόπωρο και δεύτερον, ως, όπως πάντα, έχουμε και το απαραίτητο newsletter και όσοι δεν το έχετε λάβει μπορείτε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα για να λάβετε ένα αντίγραφο και από τη συνεδρίαση του Απριλίου έχουμε τα πρακτικά θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται μέχρι το τέλο της συνεδρία, εκτός και αν υπάρξουν αντιρρήσεις. Αυτά είναι τα εισαγωγικά μου σχόλια. Κύριε Ταραμπέλα, καλώ ήλθατε. Ανέφερα την ε, σημαντική σα ε, έκθεση νωρίτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για αυτή τη συνεδρίαση. Ας ε, προχωρήσουμε τώρα στην γνωμοδότηση επίσης να καλωσορίσω τον κύριο Κρότσμαν. νομίζω ότι επανεμφανίζεται σε αυτή την επιτροπή και αναφέραμε νωρίτερα την εντολή για την έκθεσή σας ε, για την εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας υπάρχει μια αναβολή. Μήπως ε, σε ένα λεπτό μπορείτε να μας πείτε πού βρισκόμαστε. Όλοι νομίζαμε ότι θα, πέρνα, θα είχαμε μία απόφαση του Συμβουλίου, αλλά το Συμβούλιο δεν κινείται και χθε το βράδυ άκουσα ότι δεν μπορούν να αποφασίσουν τι θα γίνει. Έχουν άλλα θέματα που τους απασχολούν σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές οικολογικής αποτελεσματικότητας και δεν κινούνται επί του θέματος. Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι αν πρέπει να προχωρήσει στην Ολομέλεια και εγώ πιστεύω ότι καλύτερα θα ήταν να πιέσουμε λίγο παραπάνω, να ζητήσουμε να πάει στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο και αν δούμε τότε να κινείται το Συμβούλιο θα γίνουν οι οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις, διαφορετικά θα προχωρήσει εις ε, την Ολομέλεια το Σεπτέμβριο, έχουμε πλειοψηφία στην Επιτροπή και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και μεγάλη πλειοψηφία εις ε, την Ολομέλεια και μετά θα έχουμε τρεις μήνες να συζητήσουμε συζητήσουμε αφού τελειώσει η ε, Δανική Προεδρία ίσως καλύτερες εξελίξεις υπό την Κυπριακή Προεδρία παρόλο που λέγεται ότι η Επιτροπή επηρεάζει τις συζητήσεις διότι δεν μπορούν επαρκώς ε, να είναι εξουσιοδοτημένοι για διαπραγματεύσεις. Θα δούμε τι θα γίνει με τον εισηγητή με έναν εισηγητή και αυτή είναι η ενημέρωση που είχα να σας κάνω. Ευχαριστώ. Ε, ελπίζω ότι οι συντονιστές θα το συζητήσουν και θα μπορούσαμε να επαλέθουμε τον Ιούλιο αντί για το Σεπτέμβριο αλλά αντιλαμβάνομαι τι προτείνεται ε, ίσως να ψηφίσουμε όλο το θέμα και να περιμένουμε τι θέλουν να κάνουν οι ε, συντονιστές. Οπότε ε, περνάμε τώρα στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και με τα χαράς θα δώσω το λόγο εις την κυρία Μακλάκιν σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο κύριος Κρόιτσμαν, ο οποίος είναι εισηγητής για όλη την έκθεση, ευτυχώς είναι εδώ. Ο κύριος Παλτασάρ δεν είναι εδώ. Υπάρχει κάποιος από το ΕΛΚ, ε, δεν βλέπω κάποιον. ούτε ο κύριος Ρέπχο, η κυρία Γκέπχαρτ θα εκπροσωπήσει τους σοσιαλιστές, ο κύριος Κρόιτσμαν είναι εδώ, η κυρία Ρούλε είναι εδώ και ε, η κυρία Τζαστροζέμξκα είναι εδώ ε, εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, Οπότε, Δίνω το λόγο στην κυρία Μακλάκη να παρουσιάσει την πρόταση αυτή. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα συνάδελφοι. Το πρόγραμμα COSME έχει ως στόχο να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως στόχο να υποστηρίξει και την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 περιλαμβάνοντας όλες τις επιχειρήσεις και υποστηρίζοντας την ανάπτυξή τους. Αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Βιομηχανίας. Στόχος της γνωμοδότησής μου ήταν να επικεντρωθώ σε κάποια βασικά σημεία. Θέλω να ενθαρρύνω την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και επικεντρώθηκα ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί πολύ συχνά λέμε στην Επιτροπή μας ότι αποτελούν πραγματικά τη ράχοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρέπει οι επιχειρήσεις να δραματίσουν σημαντικό κεντρικό ρόλο σε μια Ευρώπη σημαντικής οικονομικής ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό επίση να συνειδητοποιήσουμε ότι οι επιχειρήσει συμβάλλουν πολύ στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν καλύτερε συνθήκε προκειμένου να υπάρχει ένα καλύτερο επιχειρηματικό πνεύμα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και να έχουν πραγματικά πρόσβαση στι αγορέ. Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό θα ήταν να μειωθεί το νομοθετικό άχθος, νομοθετικό φόρτος. Επίση θα πρέπει να πλουστευτεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις που μόλις τώρα ξεκινούν τη δραστηριότητά τους. Να βοηθήσουμε ουσιαστικά του πολίτες αυτού που θέλουν να στήσουν νέε επιχειρήσει θα πρέπει να καταφέρουμε μέσω του κοινοτικού αυτού προγράμματος να καταφέρουμε να δώσουμε προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και θα πρέπει να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις αυτές να καλύψουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Τα μέτρα αυτά όμως θα πρέπει να συνοδεύουν τα εθνικά μέτρα και να μην επικαλύπτουν τα υφιστάμενα εθνικά μέτρα. Οι ψηφιακές υπηρεσίες επίσης μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο. Είναι καλύτερο να καταφέρουμε να βασιστούμε στα υφιστάμενα ψηφιακά δίκτυα τα οποία υπάρχουν στα κράτη-μέλη από το να δημιουργούμε νέα δίκτυα από την αρχή. Επίση, λέω ότι είναι πολύ σημαντική η έξυπνη νομοθεσία, η ευφυή νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη αξιολόγηση των κοινοτικών μέτρων που μπορούν να συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τώρα τον τομέα του τουρισμού, συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το μέσο αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, πιστεύω ότι αποτελεί έναν από τους πολλού σημαντικούς επιχειρηματικούς τομείς και πιστεύω ότι θα πρέπει πέρα από τον τουρισμό να τονιστούν και άλλες σημαντικές υπηρεσίες και άλλοι σημαντικοί οικονομικοί τομείς όπως οι τομείς των, υπηρεσιών, των υπηρεσιών. Με συγχωρείτε. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι απαραίτητες εγγύησεις και οι πόροι που υπάρχουν στις τράπεζες προκειμένου να είναι σε θέση να χρηματοδοτούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προσβλέπω τώρα στι παρατηρήσεις των σκιωδών εισηγητών ή άλλων συναδέλφων από άλλε πολιτικές ομάδες για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα πλήρης η παρουσίαση σε αυτή και πολύ ενδιαφέρουσε και οι τροπολογίες που έχετε προτείνει. Ας κάνουμε τώρα ένα γύρο παρατηρήσεων από τους σκιώδες Ξεκινάμε με την κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ. Εγώ εκπροσωπώ τον κύριο Μήτρο Ρέπο, τον ε, εισηγητή, γιατί μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο του και έτσι δεν προλαβαίνει να είναι εγκαίρος εις ε, την ε, συνεδρίαση και επιπλέον προβλέπεται σε κάποιο άλλο σημείο αυτή η συζήτηση και είχε οργανώσει κάποια, κάποιο ραντεβού και ζητά συγγνώμη που δεν θα παραστεί σήμερα το πρωί αλλά ήθελε να μου πει ότι θεωρεί ότι η γνωμοδότηση της κυρίας Μακλάκιν είναι εξαιρετική και αξίζει να στηριχτεί αλλά ο κύριος Μέτρο θεωρεί ότι υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να τονίσει. Καταρχήν ε, το Cosme for All Program ε, και επ' αυτού θα ήθελε να τονίσει ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε μια κοινωνία η οποία γυράσκει και είναι πολύ βασικό το πρόγραμμα αυτό να εστιαστούμε όχι μόνο στις καινοτόμες ε, και ε, διεθνείς ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μάλλον μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κινούνται διεθνώς, αλλά που θα απευθύνονται συγχρόνως και σε αυτή τη νέα πελατεία. Και σχετικά με την γυράσκουσα κοινωνία θα χρειαστούμε πολύ διαφορετικές επιχειρήσεις και γι' αυτό ο εισηγητής παρακαλεί πέραν των νέων επιχειρηματιών και των γυναικών επιχειρηματιών που πρέπει να στηριχθούν να σκεφτούμε τι θα γίνει με τους μετανάστες οι οποίοι ξεκινούν επιχειρήσεις και τη μεταβίβαση μιας επιχειρήσεως από μία γενιά στην άλλη πράγμα το οποίο είναι βασικό θέμα και πρόβλημα σε μια μικρή επιχείρηση και δεύτερον πώς μπορεί να δοθεί μία δεύτερη ε, ευκαιρία σε επιχειρήσεις ε, οι οποίες ε, πτωχεύουν χωρίς να ευθύνονται αυτές αλλά οδηγήθηκαν λόγω ερήψεως ρευστότητος στην κατάσταση αυτή. Επίσης ε, είναι το πρόγραμμα COSMIC ε, ένα πολύ ευρύ πρόγραμμα που ξεπερνάει και τον ορίζοντα 2020 αλλά είναι μικρότερος ο προπολογισμός από αυτόν του, του οριζόντα 2020 οπότε πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε μπορέσουμε ε, να προσαρμόσουμε καλύτερα τα στοιχεία που έχουμε στο πρόγραμμα αυτό κατά τρόπον ώστε να υπάρχει αμοιβαία θετική αλληλεπίδραση. Και σχετικά με ε, την ε, ανταγωνιστικότητα η οποία βασίζεται στην καινοτομία θα χρειαστεί καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων όπως το κόσμο και το πρόγραμμα του ορίζοντα 2020 Όσον αφορά το πλαίσιο των προϋποθέσεων για τις επιχειρήσεις θα πρέπει ε, να βελτιωθεί και αυτό ισχύει για νέες επιχειρήσεις οι οποίες ε, πρέπει να έχουν μία καλή βάση ε, σχετικά με την ε, εξέλιξη των επιχειρήσεων ε, αυτών στις ε, διάφορες, στους διάφορους κλάδους και ιδίως στην κατάρτιση των επιχειρήσεων κάτι το οποίο θα πρέπει ίσως να εξετάσουμε πιο, πιο εκ του σύνεγγης. και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την απάντησή σας. Βλέπω ότι ήρθε και ο κύριος Μπαλτεσάρε. Αλλά καταρχήν να δώσω το λόγο στον κύριο Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ. Σαν εισηγητή του κόσμου και θα μπορώ να πω στην κυρία Γκέπχαρ ότι όλα αυτά θα αναφέρονται και ανα πάσα στιγμή μπορούμε να τα συζητήσουμε. Τηλεφωνήστε και εσείς και οι ε, σκιώδεις στο γραφείο μου να συντονιστούμε. Έχουμε και τις δικτυώσεις και τη δεύτερη ευκαιρία. Δυστυχώς όμως αυτό που που δεν μπορέσαμε είναι αντί για 2,5 δις να έχουμε 5 δις αλλά το ζητάμε ε, και το συζητάμε με τους πράσινους και τους συντηρητικούς και λέμε ότι αυτό το οποίο θέλουμε από τον ορίζοντα 2020 θέλουμε να αυξήσουμε το 0,2% σε 0,5% για να υπάρξουν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ ευρώ να αυξήσουμε και το ε, πλαφόν διότι έτσι ε, για τις μεταβιβάσεις στην ε, επόμενη γενιά οπότε δεν φτάνουν τα 150.000 ευρώ θα πρέπει να έχουμε τονίσει αυτό το επιχείρημα. Όσον αφορά την κυρία Μακλάκλιν δεν έχουμε διαφορές. Έχουμε καλύψει τον τουρισμό που επέμενε ο κύριος Ταγιάννη και όσον αφορά τις ψηφιακές παροχές υπηρεσιών τις προωθούμε αλλά δεν θέλουμε να αναφερθούμε σε ένα συγκεκριμένο τομέα όπου η ψηφιακή πτυχή είναι πολύ σημαντική. Δεν θέλουμε όμως να κατακαιρματίσουμε τους τομείς και γι' αυτό όσον αφορά την προώθηση το αναφέρετε και εσείς που είναι πολύ σημαντικό στην έκθεσή σας ε, η κατάργηση της γραφειοκρατίας επίσης και αυτό που είναι ενδιαφέρον και ε, είδα τις τελευταίες μέρες που δεν είναι σημαντικό ίσως στη Γερμανία αλλά είναι πολύ σημαντικό στη Μεγάλη Βρετανία ε, γι' αυτό και αφήσαμε το 5% διότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στα διάφορα κράτη-μέλη όταν μιλάμε λοιπόν για venture capital πρέπει να υπάρχει μία μόχλευση και είναι πολύ βασικό πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι στα venture capitals υπάρχουν και ιδιώτες και ε, ίσως κινούνται τα κεφάλαια διαφορετικά από ότι όταν πρόκειται για κρατικούς πόρους. Επίσης ε, ε, η επεξεργασία των δικτών στα κράτη-μέλη, η αξιολόγηση των επιπτώσεων, η παρακολούθηση ακολούθηση της ανταγωνιστικότητας. Χαιρετίζουμε δηλαδή όλα αυτά τα οποία εσείς αναφέρετε στην έκθεσή σας. Δεν θα υπάρξει καμία αντίφαση με αυτά μεταξύ της δικιάς σας εκθέσεως κυρίας Μακλάκλιν και της δικιάς μου και ε, ε, αν υπάρξει μία υποβολή της γνωμοδότησης της ΙΤΡΕ θα δείτε ότι όλοι συμβαδίζουμε και σας ευχαριστώ για την ε, προσοχή σας. Τέλειωσα και ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε που έχουμε τον εισηγητή στη συνεδρίαση και να είναι τόσο δεκτικό. Όμω σίγουρα και οι συνάδελφοι θα καταθέσουν και άλλε τροπολογίε. Ε, τώρα, κύριε Μπαλτασάρε, μπορείτε να απαντήσετε στην έκθεση τη κυρία Μακλάρκιν και μέρου του ΕΛΚΑ. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα την έκθεση της κυρίας Μακλάρκιν, ε, κυρίω. σε σχέση με την εξισκέψη ότι η ανάπτυξη σήμερα αποτελεί ε, προτεραιότητα ε, για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και μικρές και μεσές επιχειρήσεις αποτελούν το απαραίτητο εργαλείο, το απαραίτητο μέσο για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος. Επίσης, ε, συμφωνώ με την έμφαση που δίνεται από την εισηγήτρια στην αναγκαιότητα όχι μόνο να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις ε, και να βοηθηθούν σε αυτή τη διαδικασία διεθνοποίησης ε, και διασύνδεσης με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και με όλες τις υπόλοιπες ευκαιρίες ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς ε, μέσω εργαλείων όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο ή άλλα αλλά επίσης ε, και συμφωνώ με το ότι επαναλαμβάνει ε, το ότι πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία και ότι πρέπει να υπάρχουν λιγότερες κανονιστικές πτυχές ε, που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τον ανταγωνισμό. Όμω υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί εκ μέρους της ηγητρίας στο κείμενο που δεν με πείθουν και τόσο πολύ ή θα μπορούσα να πω ότι λείπει μια πιο διαρθρωμένη εξήγηση. Η πρώτη είναι η τροπολογία 2 που αποκλείονται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή λιγότερο από 10 υπαλλήλους σε κοινωνικέ επιχειρήσεις και βιοτεχνίες. Και θεωρώ ότι κυρίω σε ό,τι αφορά τις βιοτεχνίες, ε, τους βιοτέχνε εδώ, έχουμε μία από τις κύριες συνιστώσεις των μικρών και μέσων επιχειρήσεων που σε ορισμένες πραγματικότητες της να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του οικονομικού μας συστήματος. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ε, ότι μπορούμε να έχουμε μόνο μεγάλες επιχειρήσεις. Η διάσταση των επιχειρήσεων, ακόμη και μικρή διάσταση των επιχειρήσεων, ε, είναι θεμελιώδης για την ε, ανάπτυξη θα μπορούσαμε να δώσουμε έμφαση ε, για να δημιουργηθούν κάποια σκηνοπραξίες μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων για να μπορούν να φτάσουν στην ε, παγκόσμια αγορά. όμω το να αποκλείουμε τις μικρές επιχειρήσει, τι πολύ μικρές επιχειρήσει από αυτό το μέτρο δεν είναι κατανοητό για μένα ταυτόχρονα. Θα ήθελα να μου πει η συγγήτρια ποια λειτουργία επιφυλάσσουμε στην ενιαία θηρίδα των επιχειρήσεων, όπως την αποκαλούσαμε στο παρελθόν και που σήμερα αποδίδονται, στην οποία σήμερα αποδίδονται άλλα καθήκοντα. Αναφέρομαι στο δίκτυο Enterprise Europe. Πολύ ωραία. Αναφέρεστε επιμέρου στα διάφορα προγράμματα τη Ένωση για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Όμω η ενιαία θηρίδα είναι κάτι παραπάνω είναι κάτι πιο γενικό, αποτελεί μια συμπληρωματική υποστήριξη, μια γενική υποστήριξη που δίνεται στις επιχειρήσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξής τους, μεγέθυσής τους ε, ή ανάγκης περαιτέρω ανάπτυξης. Φυσικά, δεν ε, είναι πάγια η θέση αυτή καθορισμένη εκ των αλλά θα ήθελα να μου εξηγήσετε γιατί αποκλείεται πλήρω ο τουρισμό ε, από τι ευκαιρίε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα COSME. Ο τουρισμό σε ορισμένε χώρε ε, μπορεί να φτάνει μέχρι και στο 10% του ΕΚ αν θέλαμε πράγματι να βοηθήσουμε ή αν θέλουμε ένα κανόνα που να αφορά την Νότια Ευρώπη, παραδείγματο χάρη, αν αφήσουμε τους Έλληνες ε, εκτός τουρισμού, πώς θα τους βοηθήσουμε. Σχόλιο εκτό μικροφώνου, Όμως ε, υπάρχει μια σειρά τροπολογιών που αποκλείουν πλήρως κάθε αναφορά στον τουρισμό, και στη δημιουργία συνδέσεων, ε, πυλών, βάσεων δεδομένων ίσως ε, να δίνεται υπερβολική έμφαση σε αυτή την πτυχή στην έκθεση, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί είναι μεγάλο τμήμα του τροπολίου της εισηγήτριας, ε, όλα αυτά δεν αναφέρονται. Και τέλος, τα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα χτες και τις προηγούμενες μέρες στην Ιταλία μας δείχνουν ότι η προσοχή σε σχέση με τις καταστροφές στο βιομηχανικό κόσμο, τις συνέπειες που έχουν καταστροφές στο βιομηχανικό κόσμο, είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Και στην προηγούμενη έκθεση υπήρχε κάτι τέτοιο, ότι με περισσότερα θύματα αυτού του σεισμού στην Ιταλία, προέκυψαν ε, λόγω της κατάρρευσης κάποιων ε, εγκαταστάσεων στα εργοστάσια. Υπήρχαν εργάτες εκεί που συνέχισαν να δουλεύουν. Ίσως και η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί προτεραιότητα της ε, ανάπτυξης και την εγκέντησης και της εξοπιστίας που πρέπει να δείχνουν όλα τα συστήματα και κυρίως στα πλαίσια των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν, ε, θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις για αυτά τα θέματα. Κατά τα λοιπά, η γενική προσέγγιση με βρίσκει σύμφωνο και φυσικά πρέπει να έχουμε περισσότερους σπόρους γιατί σήμερα εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω αυτού του ταμείου. Σας ευχαριστώ. Uh, well, Ευχαριστώ για αυτά τα πολύ σημαντικά σχόλια και σας ευχαριστώ που αναφέρετε και το σεισμό στην Ιταλία. Και φυσικά τα συλληπιτήριά μας ε, και ήμουν εκεί την τελευταία φορά κάνοντας ε, κάποια έρευνα για το φάκελο ε, των μαστοκλητών και πήγαμε στην Μπολόνια για να επισκεφτούμε την Ducati και άλλες Κύριε Ρούτε, νομίζω ότι είστε τελευταία σκιώδης ε, και θα δώσω το λόγο για τους υπόλοιπους συναδέλφους αν θέλουν το λόγο. Παρακαλώ. Θα είμαι σύντομη διότι τα περισσότερα έχουν ήδη λεχθεί. Θέλω απλούστατα να τονίσω ότι η έκθεση της κυρίας Μακλάκιν κατά τη γνώμη μου είναι πολύ καλή και θέλω να τονίσω ότι συμφωνώ πλήρως με τη στρατηγική του κυρίου Κρόιτσμαν. Δηλαδή να μην αναφέρουμε συγκεκριμένα κάποιο τομέα διότι όσον αφορά τις δομές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπάρχουν τέτοιες διαφορές εντός της Ευρώπης που αν εστιαστούμε σε ορισμένους τομείς ενδέχεται να υπάρξει μία αποδυνάμωση κάποιου τομέα. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το αναφέρουμε και να είμαστε πολύ ε, πιο γενικοί. Ο τουρισμός είναι ε, βασικός για χώρες σαν την Ιταλία, αλλού είναι η κατασκευή μηχανημάτων. Ε, δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να τονίσουμε μία ε, ένα είδος επιχειρήσεων. Όπως είπε ο κύριος Μπαλταζάρε, οι μικρές επιχειρήσεις και οι ε, επιχειρήσεις μεταποίησεως είναι κάτι που θα πρέπει να στηριχθεί επίσης. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα θέλει να ε, μιλήσει πριν λάβουν το λόγο οι συγητές. Να κάνω μια-δυο παρατηρήσεις. Βλέπω καταρχάς ότι έχουμε λάβει ένα κείμενο από το Σουηδικό Κοινοβούλιο, το οποίο αντιτίθεται σε μια συγκεκριμένη πτυχή της πρότασης αυτής που έχει να κάνει με την προώθηση του εμπορίου, στο σημείο εκείνο που λέγεται ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία ουσιαστικά θα έπρεπε να διευθυντηθούν από την αρχή της επικουρικότητας όσον αφορά την προώθηση του εμπορίου. Ουσιαστικά τα όσα προβλέπονται στην νομοθετική αυτή πρόταση δεν συνάδουν με την αρχή της επικουρικότητας. Δεν ξέρω αν οι συντάκτρια γνωμοδότηση ή ο συγητής έχουν μια άποψη γι' αυτό. Κάτι ακόμα που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με την πρόταση της κυρίας Μακλάρκιν το πώς θα καταφέρουμε να θαρρύνουμε τις τράπεζες να δανείσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί αυτό που βλέπουμε πανευρωπαϊκά είναι ότι υπάρχουν πολλές τράπεζες οι οποίες προσπαθούν να βελτιώσουν τα οικονομικά τους και τον ισολογισμό τους, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι πολύ, πολύ δύσκολο πλέον για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση. Το κόστος πλέον του δανεισμού είναι πολύ μεγαλύτερο και οι τράπεζες δεν θέλουν να εκτεθούν σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες οι οποίες είναι ιδιαίτερα πιεστικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλούνται λοιπόν να βρουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και όπως λέει η κυρία Μακλάρκινγκ, ενδεχομένω θα πρέπει εδώ πέρα οι τράπεζες να συμμετέχουν περισσότερα σε κοινοτικά προγράμματα στοχευμένα για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα σύστημα παρακολούθησης και να μπορούμε να συγκρίνουμε πώ έχει κατάσταση από τη μία χώρα στην άλλη. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη πρόταση κυρία Μακλάρκιν θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Ποιο θέλει πρώτο το λόγο τώρα. Ο κύριος Κρότσμαν μάλλον πρώτος και μετά η κυρία Μακλάρκιν να συνοψίσει καταλήγοντας. Κύριε Κρότσμαν. Ευχαριστώ. Κύριε Μπαλταζάρε, όντως πρέπει να εμπλακούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, διότι στην ε, Γερμανία έχουμε πολλές ε, αυτοτελείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο τουρισμός είναι κάτι το οποίο ξεπερνά τα εθνικά όρια. Γι' αυτό ξέρω ότι ο κύριος Σταγιάννη ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Εμείς δεν αποκλείουμε τον τουρισμό αλλά δεν αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο τομέα διότι τότε θα όλοι. Εάν όμως αναφερόμαστε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βλέπουμε να υπάρχει ανάγκη δεν πρέπει να αποκλειστούν οι επιχειρήσεις αυτές. Και ιδίω αν αναφερθούμε στις ψηφιακές επιχειρήσεις πάλι υπάρχει τομεακός περιορισμός και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πιο γενικοί. Στο κόσμο ε, υπάρχει μία δυνατότητα ε, για να πούμε πώς θα υπάρξει πρόσβεση διότι στον ορίζοντα ορίζοντα 2020 είναι πολύ περίπλοκο να εμπλακεί κανείς και να συνεχίσει να περιλαμβάνεται ενώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ βασικό να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και γι' αυτό ακούσαμε ότι όταν έχουν δυσκολίες οι επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα αλλά τα καταφέρουν τότε θα επαναλάβουν την προσπάθεια αυτή και είναι βασικό αυτό και για τις Ιταλικές επιχειρήσεις και θα δούμε ότι θα υπάρξουν και άλλες αιτήσει και αυτό είναι ένα από τα μελήματά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, στείλτε μου τις παρατηρήσεις και θα δείτε ε, οι προσπάθειές μας βαίνουν προς την ίδια ε, κατεύθυνση. Ευχαριστώ και την κυρία Μακλάκη. Δεν έχουμε διαφορές και συμφωνούμε πλήρως. Μάλιστα. Πρωτού δώσω το λόγο στην κυρία Μακλάρκιν, ο κύριος Αριέσκο, θέλετε το λόγο, νομίζω ότι θέλετε να πάρετε το λόγο πριν να μιλήσετε, συγγνώμη δεν σας είχα δει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Απλώς ε, μια διευκρίνηση θέλω να κάνω. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά εγώ δεν μίλησα ποτέ για το ψηφιακό τομέα, μίλησα για την ψηφιακή αγορά. Ε, δεν θεωρώ ότι είναι τομέα ο ψηφιακό, αλλά μέσα στην ψηφιακή αγορά χωράνε όλοι οι τομεί. Έτσι λοιπόν, ήθελα να το διευκρινίσω αυτό, γιατί νομίζω ότι αποκλίνεται ο ε, ψηφιακό τομέα επειδή θεωρείται τομέα, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε εδώ για ψηφιακή αγορά. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κυρία Μακλάρκιν για να ολοκληρώσετε. Ή μήπως πρέπει να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Κομισιόν πριν να σας δώσω το λόγο για τα καταληκτικά σχόλια. Σας ζητώ συγγνώμη, γιατί είναι εδώ και εκπρόσωπο, έχουμε και εκπρόσωπο της Κομισιόν, την κυρία Τζέστρεμ Τσέσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα δώσω το λόγο στον αναπληρωτή επικεφαλή ε, της μονάδας μου. Ευχαριστώ. Άκουσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση η Κομισιόν εξέτασε το σχέδιο της έκθεσης και θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Μακλάρκιν, την εισηγήτρια, κυρίως επειδή αναγνώρισε την πολιτική σημασία ορισμένων από των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το πρόγραμμα COSME και συγκεκριμένα το, ε, σημασία την τυχόν της ε, εφιούς νομοθεσίας όπως ε, το τεστ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και, επιχειρήσεις και την εξέταση της ε, ικανότητας της αρμοδιότητας. Τώρα, να αναφερθώ σε κάποια σχόλια και να ξεκινήσω από τον τουρισμό. Η Κομισιόν δεν συμφωνεί με την πρόταση να διαγράφει η αναφορά στον τομέα του τουρισμού στον κόσμο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Ένας είναι νομικός. Ο τομέας του τουρισμού ε, έχει συγκεκριμένη νομική βάση στη Σύνθηκη της Λισαβόνας και αποτελεί μία από τις νομικές βάσεις της πρώτης κανονισμού και γι' αυτό για νομικούς λόγους η Κομισιόν έπρεπε να βάλει και αυτές τις αναφορές στον τουρισμό στους στόχους, στο αντικείμενο. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που έχουν να κάνουν περισσότερο με το ρόλο του τουριστικού τομέα, κυρίω σε περιπτώσει ε, κρίση, εποχή κρίση. Γιατί ο τομέα του τουρισμού είναι ένα από του λίγου που αναπτύσσονται, που μεγεθύνονται ακόμα και σε εποχέ κρίση. Ακόμη και τώρα, εν μέσω τη κρίση, δημιουργούνται θέσει εργασία. Έτσι λοιπόν, η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε αυτή την αναφορά στον τουρισμό και οι δράσει του τουρισμού ήδη χρηματοδοτούνται σήμερα από το πρόγραμμα Πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω σε ό,τι αφορά το δίκτυο Enterprise Europe, η Κομισιόν κατανοεί ότι κάποιες από τις τροπολογίες που εισαγάγονται θέλουν να διευκρινίσουν το ρόλο του δικτύου. Αυτό είναι πρόσδεκτο. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα με τις τροπολογίες που προτείνονται θα ήταν να περιοριστεί ο ρόλος του δικτύου, ακόμη και αν να το συγκρίνουμε με το τι κάνει σήμερα. Και νομίζω ο κύριος Μπαλτασάρ ανέφερε ορισμένες από αυτές τις στοιχές. Εμείς ως Κομισιόν πιστεύουμε ότι το δίκτυο θα πρέπει να παραμείνει η νέα θηρίδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις επιχειρήσεις One Stop Shop. Δηλαδή ε, αυτό σημαίνει ότι δεν αντικαθιστούμε, δεν αντικαθιστούμε τι γίνεται σε επίπεδο κρατομελών, αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποτελεί την ενιαία θηρίδα και θα πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω από το να δίνει έναν απλό προσανατολισμό για τα διαθέσιμα προγράμματα. Αν θέλετε να σα βοηθήσουμε να βρείτε την κατάλληλη διατύπωση, επί της συμφωνούμε ότι είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί ο ρόλο του δικτύου. Κάτι ακόμα, το σύστημα παρακολούθηση για να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν τις εγγύησεις του χρηματοδοτικού μέσου για να αυξηθεί ο δανεισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ήδη υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα που λειτουργεί υπό το τρέχον πρόγραμμα και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτό το σύστημα παρακολούθηση, όμω λεπτομερεί απαιτήσει ε, των χρηματοδοτικών μέσων παρακολούθηση ε, θα αναφέρονται με λεπτομέρειε στο χρηματοδοτικό κανονισμό που συζητείτε τώρα στα δύο όργανα στην ε, τροπολογία 24 για την ετήσια έκθεση παρακολούθηση. Η κυρία Μακλάρκιν πρότεινε να συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση αυτή και παρακολούθηση του αντικτύπου. Δυστυχώς όμως τέτοια δεδομένα συνήθως δεν διατίθεται στα τέλη του έτους, ε, κυρίως στην αρχή του προγράμματος. Προτείνει λοιπόν η Κομισιόν να έχουμε τέτοιες πληροφορίες στην έκθεση αξιολόγησης και όχι στην ετήσια έκθεση παρακολούθησης γιατί συνήθως τότε έχουμε κάποιες πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να αξιολογήσουμε και να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος του προγράμματος. Τώρα κάποιες περαιτέρω παρατηρήσεις. Θέλω να τονίσω ότι η εστίαση στους μετανάστες και σε άλλες ε, πιο δύναμες ομάδες επιχειρηματιών περιλαμβάνονται ήδη στο πεδίο εφαρμογής πρότασης και τη χάνουν χρηματοδότηση ήδη σήμερα από το σημερινό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά το διασύνδεσμο των χρηματοδοτικών μέσων μεταξύ τους για να είναι καλύτερο ο αντίκτυπο, Θέλω να τονίσω ότι το COSME και το Horizon ε, έχουν κοινή πλατφόρμα για τα χρηματοδοτικά μέσα και φυσικά η Κομισιόν ε, επιθυμεί τέτοιου είδου συνέργειε. Και τελευταίο σχόλιο, ίσως για το ότι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσει που αποτελούνται μόνο από ένα άτομο φυσικά συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα καλύπτει κάθε είδου επιχειρήσει. επικεντρώνομαστε κυρίω στι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει και εκεί περιλαμβάνονται και πολύ μικρέ επιχειρήσει. Η Κομισιόν έχει και κάποια ε, σύσσωνο σημασία παρατηρήσει για περαιτέρω τροπολογίε. Μπορούμε να τι συζητήσουμε διμερώ. Σα ευχαριστώ. Δεν αναφερθήκατε όμω καθόλου στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει με την αρχή τη επικουρικότητα, το οποίο θίγει το Κοινοβούλιο τη Σουηδία. Συμφωνείτε με την παρατήρησή του. Έχετε δίκιο. Προφανώς δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στη γνωμοδότηση του Συνδικού Κοινοβουλίου και μάλιστα έχουμε ήδη απαντήσει Νομίζω ότι υπάρχει και μια γενικότερη παρατήρηση προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επικάλυψη ανάμεσα στο εθνικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο και όσον αφορά την αρχή τη επικουρικότητα. Συμφωνεί με την προσέγγιση αυτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσον αφορά ειδικότερα τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, μέσω του προγράμματο COSME ήδη από σήμερα προσπαθούμε να κάνουμε μια χαρτογράφηση των μέτρων που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο και αυτό το οποίο θα προτείνουμε να εφαρμοστεί μέσω του προγράμματος COSME θα έχει ως αποτέλεσμα την, το πόρισμα αυτής της χαρτογράφησης. Απότερο στόχος είναι να αποφύγουμε οποιαδήποτε επικάλυψη, δηλαδή να μην έρθουμε εμείς με κοινοτικά μέτρα να αντικαταστήσουμε τα εθνικά τα οποία ήδη υπάρχουν. Θέλουμε απλώς να συμπληρώσουμε τα εφιστάμενα εθνικά μέτρα. Κύριε Μπαλτασάρε, θέλετε και εσύ... Κύριε Μπαλτασάρε, έχετε πρώτο στο λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι όσον αφορά το ζήτημα του τουρισμού τίθεται ένα ζήτημα μεθοδολογίας. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη νέα αυτή πλέον αρμοδιότητα και χρησιμοποιεί το νέο αυτό μέτρο προκειμένου να χρησιμοποιήσει κάποια νέα μέσα ανάπτυξης τουρισμού. Ενδεχομένως να μην συμφωνούμε με το ότι είναι τελικά η έκθεση αυτή το κατάλληλο όργανο προκειμένου να εισάγουμε νέα κίνητρα και νέα μέτρα, νέους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να δώσουν νέα κίνητρα για το σημαντικότατο αυτό τομέα. Θα μπορούσαμε ουσιαστικά να παραμείνουμε στον βασικό αυτό κανόνα που λέει ότι να φερόμαστε γενικότερα στις επιχειρήσεις χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην έκθεση αυτή στον τουριστικό τομέα. Ωστόσο, υφίσταται η ε, ανάγκη αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταφέρει να μεταφέρει τα νέα αυτά μέτρα σε ένα νέο νομοθετικό μέσο το οποίο θα ενισχύσει ειδικότερα τον τουρισμό. Κύριε Γκέπχαρτ, και εσείς θέλετε το λόγο και θα μιλήσει από τα κύριε Μακλάρκιν. Ε, ευχαριστώ. Προηγουμένως ε, μίλησα για τον, εν ονόματι του κυρίου Ρέπο και εδώ θα ήθελα να αναφέρω και τις προσωπικές μου απόψεις με συγχωρείτε. Ε, όπως σας είπα δεν συμφωνώ σε όλα ίσως με τον κύριο Ρέπο. Έχω μία προσωπική ερώτηση. Δεν νομίζω ότι αυτά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που μας είπε ε, είναι πλήρως ικανοποιητικά. Ε, ο τουρισμός είναι πολύ βασικός κλάδος σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και βεβαίως πολύ σωστά έτσι υπάρχει μία αρμοδιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεω για τον τουρισμό ενιαία. Αλλά ένα πρόγραμμα για προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διότι επιτέλους συμπεριελήφθη στη συνθήκη της Λισαβόνας ο τουρισμό και ότι γι' αυτό πρέπει να αναφερθεί, δεν με βρίσκει σύμφωνη. Βεβαίως ο τουρισμός πρέπει να ληφθεί υπόψη εφόσον περιλαμβάνεται στις συνθήκες αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναφέρεται ρητός σε κάποιο κείμενο σε τομείς οι οποίοι σε άλλες χώρες πέραν της Ιταλίας και της Ισπανίας είναι ίσως καλύτερο να μην αναφερθεί ο τουρισμός. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και στο πρόγραμμα αυτό όπως σας είπα αναφερθήκαμε στον κανονισμό που λέγεται πρό, ε, πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των μικρότερων επιχειρήσεων, όχι στον τομέα του τουρισμού, οπότε πρέπει να αναρωτηθώ γιατί πρέπει να υπάρχει ένας τομέας ο οποίος εκφράζεται ρητός και αναφέρεται ρητός και ε, εάν θέλουμε να προωθήσουμε τον ε, τουρισμό τότε θα πρέπει να περιλαμβάνεται και στον, στην επικεφαλίδα ένα πρόγραμμα ειδικά για τον τουρισμό αλλά ε, ή θα πρέπει όλοι να είναι ισότιμοι ή θα πρέπει να είναι ένα ειδικό πρόγραμμα διαφορετικά εγώ δεν σας καταλαβαίνω Νομίζω ότι συμφώνησε η κυρία, συμφωνούμε την κυρία ε, Γκέπχαρτ και συμφωνεί και ο κύριος Κρόιτσμαν. Η κυρία Μακλάκλιν έχει τώρα το λόγο και θα μας δώσει και το χρονικό της περιθώριο. Χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα τις συνεισφορές σας σήμερα το πρωί. Αν μπορώ να αναφερθώ στα σχόλια του κύριου Μπαλτασάρε, εγώ είχα πει ότι θα καλύψω αυτά τα σημεία στην αρχική μου παρέμβαση, όμω ε, στην ε, τροπολογία 2 ήδη περιλαμβάνονται πολύ μικρέ επιχειρήσει, όπω είπε και η Κομισιόν. Απλώ δεν ήθελα να έχω συγκεκριμένε αναφορέ ε, στι κοινωνικέ επιχειρήσει, στι βιοτεχνίε. Και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις φυσικά καλύπτονται και θα συνεχίσουν σε ό,τι αφορά την ενιαία θηρίδα, το One Stop Shop και φυσικά για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τις Επιχειρήσεις. Αυτά υφίστανται ήδη, αλλά ανησυχώ για τις επικαλύψεις σε σχέση με το τι συμβαίνει ήδη στα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν έχουμε την ενέθερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αν ήδη υπάρχει επικάλυψη, Σίγουρα έτσι δαπανάμε πόρου, παταλούμε πόρου. Έτσι λοιπόν θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν επικαλύψει και ε, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι ό,τι απορροφά τόσο κονδύλια λειτουργεί αποτελεσματικά και εξυπηρετεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεων για τον τουρισμό. Ο τουρισμό όπω και πολύ μικρές επιχειρήσεις και όλοι οι τομείς θα περιληφθούν ω μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Απλώ δεν αναφέρουμε ρητά στον τουρισμό και σε σχέση με όσο είπε η Κομισιόν. Προσπαθώ απλώς να δω πού θα ενταχθεί ο τουρισμός Δηλαδή μπορούμε να πούμε ή το, κάναμε, το βάλαμε σε αυτό το τμήμα και ίσως ε, να υπάρχουν άλλα σημεία όπου μπορεί να ταιριάζει καλύτερα και να δοθεί έμφαση εκεί. Και αυτό είναι σημαντικό, αλλά όπως είπε και η Κομισιόν, ήδη ο τουρισμός ε, είναι ένας ε, τομέας, ένας κλάδος που αναπτύσσεται και ίσως δεν χρειάζεται να δώσουμε υπερβολική έμφαση στη σημασία του ταυτόχρονα. Χαίρομαι πολύ που είναι εδώ ο κύριος Κρότσμαν ε, και έχουμε πολλές κοινέ σκέψεις για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το πρόγραμμα COSME. Ε, αναφερθήκατε στην αύξηση 5 δισεκατομμυρίων. Ε, καλή τύχη σας εύχομαι. Αλλά αν έχουμε μαζική αύξηση σε αυτόν τον προπολογισμό, θα ασφαλίσουμε ότι αυτά τα χρήματα δεν θα απορροφηθούν από το κόστο ε, τη διοίκηση, αλλά θα διοικητευτούν στην ενιαία θερίδα, γιατί πρέπει να φτάσουν στι ΜΜΕ. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, οι επιχειρήσει πρέπει να λάβουν αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ανάπτυξη και ελπίζω να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Και σα ευχαριστώ ε, για τις τροπολογίες ε, που θα στείλετε, που θα στείλετε και σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε και στους σεισμούς στην Ιταλία. Ίσως θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και σε αυτό το θέμα ρητά, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που συζητήσαμε σήμερα το πρωί που προσυπογράφουμε και θα καταλήξουμε στη συμφωνία και νομίζω ότι θα είναι πολύ ισχυρή η έκθεση που θα προκύψει από αυτή την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας, για το χρονοδιάγραμμα θα προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε και τις παρατηρήσεις κομισιών. Τώρα χρονοδιάγραμμα 7 Ιουνίου, επόμενη εβδομάδα για τις τροπολογίες και 10 Ιουλίου η ψηφορία στην ΕΜΚΟ. Σήμερα είμαι πολύ απασχολημένη. Έχω τρεις εκθέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ που ήσασταν ε, τόσο ενεργητικοί στο χειρισμό αυτού του φακέλου. Και πραγματικά αυτό μας ενδιαφέρει να έχουμε συνδυασμένες ιδέες από όλες τις επιτροπές. Ε, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Να πω και κάτι ακόμα για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Όταν αναφερόμαι σε ψηφιακές υπηρεσίες δεν το αναφέρω στο μέα. Νομίζω ότι είχατε χάθηκε στη μετάφραση. Δεν ήθελα να απομονώσω κάτι, Απλώ έλεγα ψηφιακές υπηρεσίες που μπορούμε να παράσχουμε, οι κάποια μέσα επιγραμμικά. Ήθελα να το διευκρινίσω αυτό. Ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Πρέπει να λείψω για μια σημαντική διαπραγματευτική συνεδρίαση για μισή ώρα. Έτσι, λοιπόν, στην πω καθώς ε, υπάρχει και απουσία αντιπροεδρών, θα τις αναθέσω εδώ το Προεδρία. Θα περάσουμε τώρα στη γνωμοδότηση για την Επιτροπή Προπολογισμών για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση για μας. Ο Κρίστιαν Μπουσόη είναι ο εισηγητής, ο κύριος Μπαλντασάρε είναι σκιώδης για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι εδώ. Και η κυρία Γκέπαρτ ε, ε τα έκανε όλη σήμερα το πρωί. Η κυρία Ρούλε επίσης ε, είναι διδαξιρόπιστη. Όμως ε, δεν ξέρω από τη δική μου ομάδα ποιος καλύπτει, γιατί λείπει ο αρμόδιος. Λοιπόν, ε, τώρα εφόσον όλοι είναι εδώ, να δώσω το λόγο στην κυρία Κουάιντερ για τα προεδρεύσει. Εγώ θα επανέλθω σε μισή ώρα περίπου. Κύριε Μπουζόη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Βάιλαρ. Καταρχάς να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτάσεις που έκανε για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό το οποίο έχουμε πλέον επιτάπητος είναι καλύτερο από, το, από την υφιστάμενη πρόταση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Διαβάζοντας την πρόταση αυτή εκτίμησε ιδιαίτερα την αφορά που γίνεται στην Στρατηγική Ευρώπη 2020. Είναι πολύ σημαντική, είναι κρίσιμης σημασίας. Πρέπει οι οικονομικές μας δεσμεύσεις να συνάθουν ουσιαστικά με τους πολιτικούς στόχους που θέτουμε. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό είναι ότι ακόμα και τα μέτρα αυτά δεν αρκούν. Τα συμπεράσματα της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λένε ότι ακόμα και με αύξηση 5% στο επίπεδο των πόρων σε σχέση με το επίπεδο του 2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να πετύχει όλους τους στόχους της. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πιο φιλόδοξο προπολογισμό, αλλά και μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην κατανομή των πόρων, αν πραγματικά θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους της ε, Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Βέβαια, το οικονομικό περιβάλλον δεν μας βοηθάει οι επανδιαπραγματεύσει για το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο έρχονται μια χρονική στιγμή όπου τα κράτη-μέλη διανύουν μια περίοδο οικονομική εξυγίανση. Επομένω, θα πρέπει να είμαστε κι εμεί λογικοί στι απαιτήσει μα. Εν γέννη, πιστεύω ότι θα είναι δύσκολε οι διαπραγματεύσει. Θα ήθελα τώρα πολύ σύντομα να αναφερθώ στα στοιχεία εκείνα τη πρόταση, τα οποία αφορούν ιδιαίτερα την Επιτροπή μα, εσωτερική αγορά δηλαδή και προστασία των καταναλωτών. Βρισκόμαστε στην φάση της εφαρμογής της πράξης για την ενιαία αγορά. Όλοι θέλουμε να εφαρμοστεί η πράξη αυτή και ενδεχομένω στη συνέχεια να έχουμε και μια δεύτερη τέτοια πράξη για την ενιαία αγορά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να παρέχει τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να εφαρμοστεί η πράξη αυτή. Συζητάμε βέβαια και κάποια πολιτή προγράμματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την ιστορική αγορά και του καταναλωτέ, όπω το πρόγραμμα COSME, το οποίο μόλι συζητήσαμε, το πρόγραμμα για του ε, καταναλωτέ, το πρόγραμμα για τα τελωνία και το καθεξή. Νομίζω ότι χρειάζεται μια συνεκτικότητα ανάμεσα στην εργασία που κάνουμε για τα προγράμματα αυτά και του πόρου που έχουμε στο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν πρόκειται να επαναλάβω αυτή τη στιγμή τα επιχειρήματα τα οποία ακούσαμε στην προηγούμενη συζήτηση. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι πολύ σημαντικέ για την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη. Για την πολιτική μου ομάδα και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να εφαρμοστούν και άλλες πράξεις που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις αυτές να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να υποστηρίξουμε το προτινόμενο πρόγραμμα COSME. Όπως είπαν όμως και οι συνάδελφοι, πιστεύω ότι τα χρήματα τα οποία προβλέπονται για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο δεν αρκούν προκειμένου πραγματικά να υπάρχει μια προστιθέμενη αξία. Πολύ σημαντικό είναι και το πρόγραμμα για τους καταναλωτές. Είναι πολύ σημαντικό για την προστασία των καταναλωτών. Αν θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε, να ενισχύσουμε, να πληροφορήσουμε καλύτερα τους καταναλωτές και να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους, χρειαζόμαστε πάλι ένα προπολογισμό ο οποίος να είναι στο ύψος της φιλοδοξίας του προγράμματος αυτού. Γι' αυτό προτείνω μία αύξηση στη συγκεκριμένη δημοσιονομική γραμμή η οποία συνάδει με την πρόταση που είχε κάνει άλλο συνάδελφος για το πρόγραμμα αυτό, για την έκθεση που είχαμε ιδιότερα για το πρόγραμμα αυτό προστασία των καταναλωτών. Επίση, χρειαζόμαστε του απαραίτητου πόρου προκειμένου η εσωτερική αγορά εν γέννη να λειτουργεί καλύτερα όσον αφορά του επιμέρου τομεί τη, μεταφορέ, ενέργεια κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα Connecting Europe. Θα πρέπει όμω να χρησιμοποιήσουμε και άλλου χρηματοδοτικούς πόρους, γιατί αν αρκεστούμε μόνο στο Connecting Europe δεν θα καταφέρουμε πάλι να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Οι πόροι που προβλέπονται είναι 9,1 δισεκατομμύρια για την ενέργεια, ενώ οι εκτιμήσεις τελικά δείχνουν ότι χρειαζόμαστε περίπου 200 δισεκατομμύρια, τα οποία θα πρέπει να επενδυθούν μέχρι το 2020 τα project bonds θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Είναι πολύ καλό το ότι υπάρχει εν γέννη συμφωνία προ αυτό στα κράτη-μέλη. Απλώ πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Χρειαζόμαστε να μιλάμε πλέον σε δισεκατομμύρια και όχι για εκατομμύρια. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία δεν κατάφερα να καλύψω στο σχέδιο γνωμοδότηση, όπω η φορολογία, τα τελωνία, οι επενδύσει που πρέπει να γίνουν στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Θα υποβάλω όμως κάποιε σχετικέ τροπολογίε και περιμένω τροπολογίε θα καταθέσουν και οι συναδελφοί μου και προφανώς είμαι στη θέσή σα για οποιαδήποτε άλλη πρόταση προέρθει από τους σκιώδη εισηγητές ή από άλλα μέλη της Επιτροπής μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Μπουσάη, τώρα να δώσουμε το λόγο στους εναλλακτικούς ε, Παρακαλώ κύριο Σαρίας από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Θα μιλήσω εξ ονόματος ε, του ΕΛΚ, γιατί έπρεπε να λείψει ο κύριος Μπαλτασάρε. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλό το κείμενο, συμφωνούμε. Πιστεύουμε ότι το πλέον σημαντικό είναι να βασιστούμε στην ανάπτυξη για τα επόμενα πέντε έτη και πιστεύουμε ότι είναι καλό το κονδύλι. Φυσικά δεν αρκεί, αλλά ως ένα βαθμό είναι κατάλληλο. Έτσι λοιπόν υποστηρίζουμε σε μεγάλο βαθμό ε, το κόσμο και σε όσα προτείνονται να σας πω ότι μας βρίσκεται σύμφωνους. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές κύριε Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ τον Αντώνιο Κορέα Ντεκάμπος που ε, έπρεπε να παρουσιάσει την έκθεσή του στην Επιτροπή Ήτρε και γι' αυτό δεν μπόρεσε να παραστεί εδώ. Ε, κατά τη γνώμη του πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ διότι καταρχήν ευχαριστεί τον εισηγητή για τις προτάσεις που έχει εκπονήσει και γενικώ θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό τα, οι δαπάνες που ε, καταναλώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να ε, χρησιμοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπου πραγματικά είναι προς όφελος των πολιτών. Και ακριβώς αυτό είναι στον ε, τομέα της εσωτερικής αγοράς και της προστασίας των καταναλωτών όπου υπάρχει πραγματική αποτελεσματικότητα. Λόγω της σημασίας αυτών των τομέων και των ειδικών τομέων που είναι συνδεδεμένοι με αυτού ο κύριος Κορέντε Κάμπος συμφωνεί ε, σχετικά με αυτά τα οποία λέει ο εισηγητής Μπουζόη για το πρόγραμμα των ε, καταναλωτών και την ε, νέα ανταγωνιστικότητα και το σχετικό πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και όσον αφορά το δεύτερο, έχει ως σχόλιο ότι η μεγαλύτερη δυσκολία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή είναι η δυσκολία να μπορέσουν να έχουν πιστώσεις και οικονομική ε, στήριξη δηλαδή όχι τόσο πολύ η δυνατότητα να αναπτυχθούν ε, επιχειρησιακά αλλά η έλλειψη πιστώσεων και αυτό δύο στις χώρες που είναι πιο αδύναμες οικονομικά αυτή την εποχή. Εξού και εδώ θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινητοποιηθεί και να βοηθήσει περισσότερο κατά τρόπον ώστε να ε, μπορέσει να ε, βελτιώσει το κλίμα στα κράτη αυτά για αυτόν τον τομέα. Επίσης λέγει ότι είναι κρίμα ότι οι πόροι που προβλέπονται είναι τόσο περιορισμένοι με 340 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και ότι έτσι δεν μπορεί το πρόγραμμα αυτό να έχει πραγματικά μεγάλη επίδραση αλλά είναι πολύ θετικό αυτό το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή η απλοποίηση των διαδικασιών και οι δυνατότητες συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, σε ε, χρηματοοικονομικά ε, μέσα και προγράμματα. Ο σκιώδης εισηγητής είναι βέβαιος ότι ε, θα έχει μία καλή συνεργασία με τον κύριο Μπουζόη και ότι θα υπάρξει ευρεία συνένεση σχετικά με τις ε, ε, δικές μας ανησυχίες για να τις παρουσιάσουμε στην, στην, επιτροπή η οποία έχει αναλάβει το θέμα. Η κυρία Ρούλε και εγώ ε, πρέπει να στηρίξω τον κύριο Μπουζόη και να σας πω ότι η δικιά μας συμμετοχή σε αυτό το θέμα σαν επιτροπή είναι περιορισμένο. Πρέπει όμως να δούμε πώς θα υπεραμεινθούμε των συμφερόντων μας έναντι των άλλων επιτροπών. Ευχαριστώ. Η ECR τώρα έχει εκπρόσωπο, η συντηρητική. Ε, όχι, ούτε η Γκουε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η έκθεση είναι αδιαμφισβήτητη, ούτε η, η έχουν εκπρόσωπο. Ε, πρόσωπος της Επιτροπής δεν υπάρχει και πριν δώσω στον κύριο Μπουζόη το λόγο για να δευτερολογήσει έχω μία ερώτηση. Άκουσα από τα σχόλια ότι ο όγκος της χρηματοδοτήσεως είναι περιορισμένος. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει ε, εάν έχουμε ε, τόσο περιορισμένο μέσα να συνδυάσουμε και την οδηγία για την διακίνηση των πληρωμών Λοιπόν για να βελτιωθούν οι δυνατότητες χρηματοδοτήσεως για να κινούνται πιο γρήγορα τα εμβάσματα είναι κάτι το οποίο είχαμε στηρίξει και πέρυσι. Οπότε έχει όντως εφαρμοστεί το θέμα αυτό σε διάφορα κράτη όπου δεν είχε προχωρήσει. Ίσως η Επιτροπή θα μπορούσε επί του θέματος να μας απαντήσει, αν όχι σήμερα, στη συνέχεια τηλεφωνικά για να μας πει πόσο έχει προχωρήσει η εφαρμογή αυτή της οδηγίας Κύριε Μπουζόη. Λοιπόν, ε, τότε θα μιλήσετε κι εσείς πριν ε, δευτερολογήσει ο κύριος Μπουζόη. Πρόεδρε, πριν μιλήσω εξονόματος τη ομάδα, ε, τώρα θα να μιλήσω ω συντονιστή της ομάδας εργασίας ηλεκτρονικού εμπορίου. Να αναφέρω στο σημείο 5. Γίνεται λόγο για την ενιαία αγορά ενέργεια και για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Εγώ νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία, καθώ ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε είναι το πρόβλημα της ανεργία. Και ξέρετε ότι πρόκειται για δύο τομές που πρέπει να εκμεταλλευτούμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σίγουρα στην ψηφιακή αγορά. Όπου εγώ θα μπορούσα να συνεισφέρω περισσότερο. Πρόκειται για ένα σημείο, πρόκειται για ένα τομέα όπου έχει υπάρχει μεγάλη δυναμική για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Και όλοι ξέρουμε ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, δημιουργούν θέσει εργασία, όχι μόνο μεγέθυνση. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό που αναφέρεται αυτό στο σημείο 5 και θέλω λοιπόν ε, να χαιρετήσω αυτή την αναφορά στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Ο κύριος Μπουσόη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, που είπαν καλά λόγια για την πρότασή μου. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Ρέση Τσεβερία. Συμφωνώ ότι είναι ανεπαρκής ο προπολογισμό, αν και είναι κατάλληλος. Θα προσπαθήσουμε να ζητήσουμε περισσότερους πόρους και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά με την, εσωτερική αγορά, με την πολιτική εσωτερικής αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Κατανοούμε ότι σε ορισμένα κρατημέλη υπάρχουν οικονομικέ δυσκολίε και γενικά το πολιτικό κλίμα στην Ευρώπη δεν είναι πάρα πολύ θετικό για την αύξηση των ευρωπαϊκών προπολογισμών. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλο, Αλλά θα προσπαθήσουμε να ζητήσουμε περισσότερου πόρου. Και καθώ πιστεύω ότι η ενιαία αγορά ενέργεια και η ψηφιακή ενιαία αγορά είναι επίση ε, καθοριστική σημασία για το μέλλον μα. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Γκέπχαρτ Συμφωνώ ότι θα πρέπει να δαπανούμε πιο αποτελεσματικά τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συμφωνώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις ΜΜΕ είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η δυσκολία δανοδότησης. Και εδώ το θέτω ως πρώτη προτεραιότητα για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Το κόσμο δεν αρκεί, θα πρέπει να βρούμε και άλλες λύσεις. Ευχαριστώ και την κυρία Ρούλα για την υποστήριξή της και φυσικά περιμένω και τη συνεισφορά των πρασίνων για τις προτάσεις μου. Και για να απαντήσω και στην κυρία Βάιλερ, προσπαθούμε και δύο να συμμετέχουμε στην ε, μεταφορά στην ιστορική νομοθεσία με σωστό και ταχύ τρόπο της οδηγίας για τις καθυστερημένες πληρωμές. Καλό είναι να, θέτουμε, να θέσουμε κάποια ερώτηση στην Κομισιόν και να ζητήσουμε μια εξήγηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια συνολική έκθεση. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τη Ρουμανία, για τη χώρα μου, όπου δυστυχώς ε, δεν έχουν γίνει και δεν έχει σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδο για τη μεταφορά αυτή τη οδηγία στην εσωτερική νομοθεσία και πιστεύω ότι και άλλε χώρε που είχαν προβλήματα με αυτέ τι καθυστερημένε πληρωμέ δεν έχουν σημειώσει πρόοδο μέχρι τώρα. Φυσικά έχουν ακόμη λίγο χρόνο μέχρι τα τέλη του έτους. Αλλά όπως είπατε και εσείς, πιστεύω ότι το να αποφύγουμε τις καθυστερημένες πληρωμές θα μπορούσε να βοηθήσει και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ε, προκειμένου να υπάρχει ορθή ροή των πληρωμών. Προτείνω το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 18 Ιουνίου, το 12 μεσημέρι και προτείνω ψηφοφορία να λάβει χώρα σε αυτή την Επιτροπή στις 10 Ιουλίου, δηλαδή πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank, Herr Ευχαριστώ κύριε Μπουζόη. Και τώρα έρχομαι στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 18 Ιουνίου. Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι οι διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και η κατάργηση της απόφασης. Η κυρία Καλνάιτε είναι εδώ και ε, μου ελέγχθη ότι έχουμε φροντίσει να υπάρχει διερμηνία από τη γλώσσα της για να δούμε αν είναι οι υπόλοιποι εδώ. Ο κύριος Σίβιτς για τους σοσιαλιστές δεν είναι εδώ. Η κυρία Γκέπχαρτ θα τον αντικαταστήσει. Για τους φιλελεύθερους ο κύριος Μπουζόη. Η κυρία Ρούλε για τους πράσινους. Να και ο κύριος Σίβιτς. Για την ECR ο κύριος Βίλαν που δεν έχει έρθει ακόμη. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και η κυρία Καλνάιτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Πραγματικό επίτευγμα αυτό στην Επιτροπή μας, πρέπει να το πω. θα αναφερθώ στην ε, γνωμοδότηση αυτή που έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές συνεργειακές υποδομές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδης ηγητές από τις ε, άλλες πολιτικές ομάδες για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και για τις προτάσεις που υπέβαλαν. Να ευχαριστήσω επίσης όλους τους συμβούλους καθώς επίσης και το προσωπικό της γραμματείας που συνέβαλαν και αυτοί πολύ με την εργασία τους και είμαστε πλέον ε, σε θέση να ψηφίσουμε αύριο στην Επιτροπή μας για την γνωμοδότηση αυτή. 17 τροπολογίες συνολικά κατατέθησαν, εκ των οποίων οι περισσότερες ενσωματώθηκαν, τουλάχιστον προσπάθησαν να τις ενσωματώσω στο κείμενο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να στηρίξουμε όλες τις τροπολογίες που λάβαμε. Και αυτό γιατί εν μέρη δεν είχαν να κάνουν με την αρμοδιότητα της Επιτροπής μας ή σε άλλες περιπτώσεις ερχόντουσαν σε αντίφαση με την πολιτική κατανόηση που είχα εγώ και οι δισυγιτές για το υποεξέταση ζήτημα. Πρέπει να σας πω ότι καταφέραμε να καταλήξουμε τελικά σε μια ισορροπημένη γνωμοδότηση μια γνωμοδότηση που έχει να κάνει με την εντολή που, έδωσε, που δόθηκε στην Επιτροπή μας να γνωμοδοτήσει, έχει να κάνει με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες Επιτροπής μας και πιστεύω ότι θα συμβάλλει σε μια καλύτερη αποτελεσματικότητα της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Παράλληλα θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει στα πλαίσια της συνθήκης. θα πρέπει να καταφέρουμε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές από τις αλλαγές που επέρχονται στις τιμές. Έχω υποβάλει μια σχετική τροπολογία και έλαβα και άλλες τροπολογίες στη συνέχεια, οι οποίες βοηθούν ουσιαστικά στο να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Θα πρέπει να έχουμε σταθερές τιμές καταναλωτή θα πρέπει οι λογαριασμοί που φτάνουν στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην παρουσιάζουν αυξήσεις. Ενισχύσαμε επίσης την ενεργειακή ασφάλεια. Είναι και αυτό μια σημαντική συμβολή στην γνωμοδότησή μας και, σε μια, και έχει, να κάνει, έχει σχέση με μια γνωμοδότηση που είχαμε υποβάλει το 2009 στα πλαίσια της Επιτροπής μας. Το πρόγραμμα Connecting Europe, συνδέοντας την Ευρώπη, το μέσο μάλλον αυτό, είναι ένα σημαντικό μέσο το οποίο θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλλει στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μεγαλύτερες επενδύσεις σε κάποιες βασικές ενεργειακές υποδομές, οι οποίες με τη σειρά τους θα αυξήσουν την εσωτερική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίοδο οικονομικής κρίσης την οποία διανύουμε. Συζητώντας με τους συναδέλφους το κείμενο αυτό, πολλές φορές αναφερθήκαμε και στο ζήτημα της μεθοριακής συνεργασίας. Πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή που έχουμε την ενεργειακή στις μεθοριακές ζώνες της Ευρώπης. Υπάρχουν ορισμένα μέσα τα οποία αναφέρονται και τα οποία θα μπορούσαν να ισχύσουν την διασυνεριακή συνεργασία και τα οποία τα αναφέρουμε και τα τονίζουμε στην γνωμοδότησή μας. Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Κορέρα Τεκάμπος, ο οποίος είναι ο βασικός εισηγητής στην Επιτροπή Ήτρε για τον κανονισμό αυτό. Συνεργαστήκαμε λοιπόν μαζί προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, προκειμένου να έχουμε μια μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό και προκειμένου να προωθήσουμε νέες ενεργειακές πηγές. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και μία αμοιβαία ολοκλήρωση των ενεργειακών υποδομών και δικτύων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Καρνάιτε. Τώρα ο λόγος στους εισηγητές και καταρχήν από τους ε, σοσιαλδημοκράτες ο κύριος Μάρεκ ε, Τσίβιτς. Ευχαριστώ. Είμαστε κοντά στην τελική ε, ευθεία και είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένως. Τώρα έχουμε 17 τροπολογίες και πρέπει να σας πω ότι οι τροπολογίες αυτές συνοψίζουν τη συζήτηση αυτή και αποτελούν ε, μία περίληψη της συζήτησης. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει δυνατότητα δεν νομίζω ότι θα κάνουν κακό ή στην έκθεση διότι πιστεύουμε ότι όλα αυτά έχουν σχέση με τα συμφέροντά μας και η προστασία των καταναλωτών πρέπει να αναφέρεται χωρίς να είναι το επίκεντρο αυτού του ψηφίσματος το οποίο είναι ένα πολύ πιο τεχνικό και πολιτικό έγγραφο και εν μέρη πρόκειται και για ένα δημοσιονομικό έγγραφο. Οπότε όλα αυτά τα οποία έπρεπε να τονιστούν έχουν περιληφθεί και τώρα μεταξύ σοσιαλιστών θα συζητήσουμε ε, τον κατάλογο ψηφοφορίες. Δεν περιμένω ούτε εκπλήξεις ούτε και διαφωνίες αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει αυτή η δημοσιονομική πτυχή που δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα αλλά είναι το θέμα των ε, σχέσεων των πόρων αυτών που προέρχονται από το Ταμείο Συνοχής και αυτό δεν αφορά τη δικιά μας Επιτροπή. Θα πρέπει να συζητηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι οποίοι μας είπαν ότι υπάρχει Υπάρχει μία πολύ σημαντική πρόκληση που μας περιμένει σχετικά με την ενέργεια και θέλω να σας πω ότι οι διαφορές στις ενεργειακές τιμές κυμαίνονται στο 30% σε ορισμένες περιοχές. Οπότε εάν υπάρξουν αυτά τα ενεργειακά δίκτυα τα οποία θα είναι πιο ολοκληρωμένα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ε, ενιαίας αγοράς ε, που θα είναι και η απάντησή μας στην κρίση και γι' αυτό ελπίζω ότι πριν την ψηφοφορία θα έχουμε καταλήξει και θέλω ε, να ευχαριστήσω την κυρία Καλνάιτε την εισηγήτρια για την πολύ ε, επαγγελματική αντιμετώπιση της και ε, ιδίω την κατανόηση για εισηγητές σαν εμένα που δεν ακολούθησαν τη γραμμή και να ευχαριστήσω και πάλι για όλη τη συνεργασία Ευχαριστώ. Η κυρία Ρούλε για τους πράσινους τώρα. Λοιπόν, και εγώ μπορεί να είμαι σύντομη διότι η συνεργασία με την εισηγήτρια ήταν καλή και την ευχαριστώ για την καλή έκθεση αλλά για ορισμένες τροπολογίες έχω προβλήματα και δεν είναι εδώ ο κύριος Σμιτ του οποίου οι τροπολογίες με προβληματίζουν ε, γιατί ζητά κατάργηση ε, που δεν είναι αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής οπότε τότε Οπότε θα έπρεπε να συζητήσουμε και την αποτελεσματικότητα της ενεργείας και ε, τον ε, περιορισμό της ενεργείας. Πράγμα που δεν είναι της αρμοδιότητάς μας και δεν μπορούμε να συζητήσουμε εδώ. Αυτό που είναι αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής είναι η Επιτροπή για τους καταναλωτές ε, και τα υπόλοιπα θέματα πρέπει να συζητηθούν στην Επιτροπή Ήτρε. Ευχαριστώ κυρία Ρούλε. Ο επόμενος εισηγητής είναι ο κύριος Άνταμ Μπίλαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία εισηγήτρια. Πιστεύω ότι εργαστήκατε πάρα πολύ σκληρά για τις εκθέσεις και για, τις, ε, για την έκθεση και για τις τροπολογίες και νομίζω ότι είναι πολύ ισορροπημένη η εκθέση αυτή και δεν προς σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τις ε, ε, ενεργειακές υποδομές για την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν υποστηρίζω την έκθεση κυρία Καλινέτη. Νομίζω ότι η εφαρμογή αυτού του εγγράφου θα είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη των ε, στόχων και νομίζω ότι από τη δική μας Επιτροπή θα πρέπει να δοθεί έμφαση ότι θα πρέπει να οδηγήσει σε δραματική αύξηση στις τιμές της ενέργειας για το μεσονικό κυριό. Νομίζω ότι η ανάπτυξη του τομέα τη ενέργεια είναι πολύ σημαντική για την ενιαία αγορά. Το αναφέραμε και στο παρελθόν επίση για την ανάπτυξη των επιχειρησιών μα, κυρίω ε, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί για αυτέ οποιαδήποτε αύξηση τιμέ ε, θα μεταφραστεί σε μεγάλε οικονομικέ δυσκολίε. Όταν ε, μιλάμε για τα έργα που είναι τα πιο σημαντικά, τα project τα πιο σημαντικά, θα πρέπει να επιλέξουμε αυτά που δεν παραβιάζουν την αρχή τη ανταγωνιστικότητα και επίσης ε, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι στρατηγικές λύσεις για την οικονομία μας. Εγώ υποστηρίζω τις περισσότερες από τις τροπολογίες που προτείνονται, κυρίως ό,τι αφορά τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Η ομάδα μου θα υπερψηφίσει τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπίλαν. Υπάρχουν άλλοι που ζητούν το λόγο. Ο συνάδελφοι, ο κύριος Μπουζόη, έχετε το λόγο, με συγχωρείτε, δεν σας είχα δει. Θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρους του κύριου Σμίτ που είναι σκιώδης μας. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη συμβαστική της προσέγγιση. Οι φιλελεύθεροι υποστηρίζουν τις περισσότερες τροπολογίες αλλά και τις συμβαστικές τροπολογίες. Ε, ο συνάδελφος ο Σκιώδης από το ΑΛΤΕ έχει κάνει μια αναφορά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ε, το να είναι χαμηλές οι τιμές ε, στην ενέργεια είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό αφορά και τις ΜΜΕ και τους καταναλωτές. Θέλουμε να υπάρχει ομαλή λειτουργία των έργων και να υπάρχει διασυνοριακή ε, συνεργασία στον τομέα TEN-E ε, των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα πρέπει να επιφέρουν την ε, ευρωπαϊκή αξία και διασυνοριακή διάσταση είναι πολύ σημαντική στον τομέα αυτό, καθώς και η ευθύνη των κρατών μελών είναι να παρουσιάσουν ωφέλη για τους πολίτες και να καλύψουν τα κενά αναφέρονται και κάποιοι κίνδυνοι. Υπάρχει ο κίνδυνος να μπερδευτούν οι ε, αρμοδιότητες των κρατών μελών με τις αρμοδιότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως ε, θεωρούμε ότι η συγκήτρια έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και θα ψηφίσουμε σε επί μια ισορροπημένη εκδοχή της γνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να καλέσω προσυζήτηση τον ο, ε, ο, διευθυντή της ΕΝΑ ο οποίος θα μπορούσε να μας διαφωτίσει σε διάφορα θέματα ε, ιδίω σχετικά με τη σιωπή και την αδράνεια που υπάρχει σε ορισμένα κράτη-μέλη ε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση κάθε φορά που έρχομαι στην Επιτροπή σας, γιατί κάθε φορά μου δίνει τη δυνατότητα να συζητώ μαζί σας και να εξηγώ κάποια πράγματα. Μόλις ήρθα από την Ήτρε που μου δώσανε μόνο πέντε λεπτά για να αφαιρθώ σε μια έκθεση που είχε 850 τροπολογίες. Αυτό για να σας ενημερώσω λίγο για το πώς έχουν τα πράγματα σε κάποιες άλλες επιτροπές. Χάρηκα πάρα πολύ όταν ήμουν ήδη παρόν εδώ τον Απρίλιο που κάνετε την πρώτη συζήτηση και είχα τη δυνατότητα τότε να απαντήσω και σε κάποιες ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής σας. Η εργασία της κυρίας Καλνιέτε, της Επιτροπής, της Συγκεκριάς, με συγχωρείτε, είναι πολύ καλή. Όλα κινούνται ουσιαστικά στο δρόμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προς τους στόχους που είναι κοινοί για όλους μας, νομίζω. Το να καταλήξουμε δηλαδή σε πραγματικές διευρωπαϊκές συνεργειακές υποδομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση πράγμα το οποίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στον ενεργειακό εφοδιασμό για όλους τους πολίτες, βασιζόμενοι σε μια μεγαλύτερη ποικιλία και διαφορετικότητα ενεργειακών πηγών. Ξέρετε ότι θέλετε να μειώσουμε το ποσοστό άνθρακα και ορυκτών καυσίμων στον τομέα της ενέργειας στην Ευρώπη. Τα όσα λοιπόν συζητάμε εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικά. Τα αναφέρατε όλα αυτά και είπατε επίση ότι είναι πολύ σημαντικό να εργαστούμε και προ όφελο του καταναλωτή. Όντω, αυτό αληθεύει. Πολύ συχνά δεν δίνουμε την απαραίτητη σημασία στον καταναλωτή και ο καταναλωτή δεν αποφελείται επαρκώ από το άνοιγμα τη ενεργειακή αγορά. Το εξήγησα και την προηγούμενη φορά, είναι πολύ σημαντικό πάντω να το έχουμε κατά νου, ότι κάθε φορά που μιλάμε για υποδομές μετακίνησης της ενέργειας, φυσικής ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, ενέργειας φυσικού αερίου, με συγχωρείτε, είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι ε, ε, δεν θα πρέπει να α, ε, επιβαρύνεται ιδιαίτερα ο τελικός καταναλωτής από τον λογαριασμό ο οποίος φτάνει σε αυτόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε τις υποδομές αυτές προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές για τον καταναλωτή. Αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές προκειμένου να διαχέεται σωστά ηλεκτρική ενέργεια το φυσικό αέριο προς τον καταναλωτή, τότε ο καταναλωτής θα εξαρτάται ιδιαίτερα από μια εθνική αγορά, η οποία ενδεχομένω με τη σειρά τη να εξαρτάται ιδιαίτερα από συγκεκριμένου πόρου ή από ένα εξωτερικό προμηθευτή, και αυτό με τη σειρά του επηρεάζει ιδιαίτερα τι τελικέ τιμέ. Το να καταφέρουμε να διασυνδέσουμε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενό διευρωπαϊκού δικτύου φυσικού αερίου, για παράδειγμα, το οποίο θα καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη, και που θα επωφελείται πολλών διαφορετικών πηγών φυσικού αερίου, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωφέλιμο για τον καταναλωτή, καθότι δημιουργεί προσιτές τιμές. Τώρα για την ηλεκτρική ενέργεια. Ξέρετε ότι χρησιμοποιούμε την ηλική ενέργεια εκεί πέρα που υπάρχει ήλιος ή την νεολική ενέργεια εκεί πέρα που υπάρχει άνεμος ουσιαστικά έχουμε εναλλακτικέ πηγέ ηλεκτρική ενέργεια εκεί πέρα που δεν βρίσκεται ουσιαστικά ο καταναλωτή. Είναι πολύ σημαντικό η παραγόμενη κατά αυτόν τον τρόπο ηλεκτρική ενέργεια να μεταφέρεται μετά στον καταναλωτή. Αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε το στόχο του 20% μέχρι το 2020 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο energy mix το οποίο ακολουθούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε αυτές τις ενεργειακές υποδομές προκειμένου να γίνεται σωστά η μεταφορά της ενέργειας. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και είναι πολύ σημαντικά και για τον καταναλωτή βέβαια. Και νομίζω ότι αυτό το έχετε καταλάβει εσείς πάρα πολύ καλά και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ε, υποστήριξή σας, ε, όπως αυτή ε, αντανακλάται στην έκθεση της κυρίας Καλιέντε, αλλά και στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν χρησιμοποίησατε την ε, πιθανότητα και τη δυνατότητα που είχατε να αναπτύξετε περισσότερο εδώ αυτά τα οποία δεν μπορούσατε να ε, αναπτύξετε στην Επιτροπή Ήτρε. Αλλά υπάρχει και ο εισηγητής της Ήτρε εδώ. Θέλετε να μας πείτε πώς έγινε η συζήτηση στην Ήτρε κύριε Βίλαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόλις ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην Ήτρα, σε γενικέ γραμμές, η πρότασή μας ε, ουσιαστικά συνάδει με την πρόταση της Κομισιόν, όμως ε, καθιστά κάπως ε, πιο διαφανή τα πράγματα. Τα σχόλια γενικά ήταν πάρα πολύ θετικά σε σχέση με τις τροπολογίες. Εν τω μεταξύ, θέλω να τονίσω δύο τεινά. Το πρώτο έχει να κάνει με την πρόταση των φιλελευθέρων να αποσυρθεί πλήρως το άρθρο 15 από την πρόταση αυτή με το επιχείρημα ότι πρόκειται για οικονομικά θέματα και όλα τα οικονομικά θέματα θα πρέπει ε, σωρευτικά να παρουσιαστούν στο μέσο διαστήμησης για την Ευρώπη, Correct Europe Facility, και σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες νομοθεσίες ε, για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών μεταφορών κτλ. Και, και υπάρχει και ένα άλλο σχόλιο, ένα άλλο σύνολο σχολείων από τους βουλευτές που είναι το εξή. Υπερασπίζουν το θέμα της επιστροφής στην ενεργειακή αυτάρκεια ορισμένων χωρών. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι υπέρ της Ένωσης. Πολλοί συνάδελφοι και από το ΕΛΚ ε, είναι στην πλευρά μας. Η Κομισιόν ε, είναι μαζί μας κατά της διαγραφής ε, του άρθρου 15 γιατί καταρχήν ε, υπάρχει νομικό πρόβλημα, δηλαδή το άρθρο αυτό είναι ουσιαστικής ε, σημασίας. Ε, στο άρθρο αυτό έχουμε τα κριτηρία ταξινόμησης και παραπέμπει ουσιαστικά στο σχετικό παράρτημα το άρθρο αυτό και χωρίς το άρθρο αυτό υπάρχει ουσιαστικά θα έχουμε ένα, ένα λιπές αποτέλεσμα για να ξέρουμε ποιο είναι το ποσό που εκτεμιεύεται για τα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, ε, για να οριστούν κατόπιν τα κριτήρια. Εγώ νομίζω ότι ακριβώς εδώ έχουμε το αντίθετο επιχείρημα, δηλαδή ε, εμείς ε, θέλουμε να καθορίσουμε κριτήρια δεν είναι ε, να αντιμετωπίσουμε επιμέρους προβλήματα, πρέπει όμως να καθαρίσουμε τα κριτήρια και να ασκήσουμε πίεση έτσι ώστε να είναι εξαντλητικά τα κριτήρια αυτά, να είναι πολύ συγκεκριμένα, να πάνε εις βάθος, αλλά πρέπει να είναι γενικά και αφηρημένα, όπως πρέπει να είναι πάσα νομοθεσία. Και κατόπιν η εφαρμογή θα γίνει από τα αρμόδια όργανα, από τα εκτελεστικά, δηλαδή από Κομισιόν και Συμβούλιο. Τώρα, ε, το να λέμε εδώ ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο αν ε, αρχίσουμε τώρα να καθορίζουμε τα κριτήρια πριν έχουμε τα χρήματα, νομίζω ότι είναι ακριβώ το αντίθετο από αυτό που τελικά θέλουμε να κάνουμε και επιδιώκουμε να κάνουμε. Η πρόταση αυτή, μάλλον η θέση αυτή, ήταν μειοψηφική στην Επιτροπή Ήτρα. Και σε γενικέ γραμμέ, θεωρώ ότι έχουμε μάλλον πάρα πολλέ τροπολογίε, 845-846, αλλά νομίζω ότι μπορεί να εγκριθεί η έκθεση αυτή, πιθανότατα θα αναβληθεί η ψηφοφορία στην Επιτροπή Ήτρε για τον Ιούλιο. Όμως πιστεύω ότι ξεκολουθούμε να διατηρούμε την προθεσμία για να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις το Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κορέρα για τη σύντομα ενημέρωση του τι γίνεται στη γειτονική ε, επιτροπή και αν δεν υπάρχει κανείς άλλος που ζητά τον λόγο θα δευτερολογήσει η κυρία Καλνέιτε αν θέλει να πει κάτι και να συνοψίσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν Ευχαριστώ και τους ομιλητές από τις υπόλοιπε πολιτικές ομάδες για τα ευγενικά τους λόγια. Πιστεύω ότι έχουμε προετοιμαστεί καλά για την ευρύνη ψηφοφορία. Η γνωμοδότηση θα υιοθετηθεί. ξέρετε, μας είπε η κυρία Ρουλό σχέση Ρούλε, σχετικά με τις προσθήκες του κυρίου Σμιτ. Όμως ε, το ΕΛΚ θα τις υποστηρίξει. Και πάλι Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κορέντε Κάμπος για την πολύ καλή δουλειά του στην Επιτροπή Ήτρε και τον Ιούλιο στην Ολομέλεια. Όλοι θα ψηφίσουμε την εκθέση αυτή. Σας ευχαριστώ. Gut, vielen Dank. Damit ist die Debatte zum Bericht Ευχαριστώ. Έτσι έκλεισε η συζήτηση αυτή. Αύριο το πρωί θα ψηφίσουμε και πιστεύω ότι τώρα έχουμε μισή ώρα διάλειμμα καφέ και δεν ε, θα προχωρήσουμε κατευθείαν διότι στη συνέχεια έχουμε μια κοινή επιτροπή με την επιτροπή ε, ε, μια κοινή συνεδρίαση με την επιτροπή μεταφορών την οποία έχουμε προβλέψει για τις 11 ε, μας προσκάλεσαν ε, χθες ε, οπότε τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών οπότε νομίζω μέχρι τις 11 παρα 5 καλό θα ήταν να κάνουμε ένα διάλειμμα για καφέ ή τέλος πάντων ό,τι θέλει ο καθένας.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 Uh, so uh, can uh, members of the Transport Committee Να καλωσορίσω και τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών στην κοινή αυτή συνεδρίαση, στην δεύτερη που κάνουμε όσον αφορά το e-call, την υπηρεσία e-call. Χαίρομαι πολύ που μπορούμε να οργανώσουμε εμεί αυτή τη φορά τη συνεδρίαση. Αυτή την προηγούμενη φορά η κοινή συνεδρίαση είχε γίνει στην Επιτροπή Μεταφορών. Να καλωσορίσω επίση και τον Ντομίνικ Κρικέ, ο οποίο είναι εδώ πέρα από την Επιτροπή Μεταφορών, και την, τον κύριο Κόχ και την κυρία Σάνλοβαν, του δύο συγητέ από τι δύο επιτροπέ. Θα ήθελα να καλωσορίσω θα συζητήσουμε τον μεγάλο αριθμό τροπολογιών, 150 τροπολογίες συνολικά που έχουμε λάβει για την πρόταση αυτή, οι οποίες καταδεικνύουν το γενικότερο ενδιαφέρον για αυτή την πρόταση. Έχουμε επίσης και σκιώδεις συγητές και από τις δύο επιτροπές. Σε λίγο θα ζητήσω από τον κύριο Κόχ, τον ε, εισηγητή από την Επιτροπή Μεταφορών, να ξεκινήσει τη συζήτηση. Θα ακούσουμε την κυρία Σεχαλνοβά στη συνέχεια. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τον α, ε, εκπρόσωπο του ΕΛΚΑ, του Νουν Από τους φιλελεύθερους, ε, ο κύριος Μπένιαν έχει φτάσει πολύ ωραία. Σας καλωσορίζουμε. Ο Φιλ Μπένιον λοιπόν έχει έρθει εκπροσωπώντας τους φιλελεύθερους. Μπορείτε να καθίσετε εδώ μπροστά. Και μία κάρτα θα σας δώσουμε. Η κυρία Ρούλη, επίσης είναι από τους Πρασίνους. Ο κύριος Τέιλορ δεν τον βλέπω. Α, είναι εδώ. κύριος Τέιλορ είναι στην αίθουσα και εγώ εκπροσωπώ την ομάδα μου. Κυρία Ρόσμπαχ δεν νομίζω ότι έχει έρθει. Ο κύριος Ντε Ιόγκ, δεν ξέρω. κυρία Φώστερ είναι εδώ μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πιστεύω. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε αμέσως στη συζήτηση των τροπολογιών θα καλέσω κάθε ένα από τους ηγητές να αναφερθεί στις τροπολογίες και στη συνέχεια θα ακούσουμε τους σκιώδεις ηγητές και οποιονδήποτε άλλο στη συνέχεια θέλει να πάρει το λόγο. Να καλωσορίσω επίσης την ομάδα από τρεις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται με την έκθεση αυτή. Έχουμε εκπρόσωπο από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας, τον κύριο Στον Μέσ, όχι, από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών ποιο είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς. Ο κύριο Σολ Μάσατζιτς είναι εδώ και ο κύριο Νταβίλα από την Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας. Θα έχετε και εσεί χρόνο προκειμένου να παρουσιάσετε την άποψή σα. Πολύ ωραία. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Κύριε Κόχο. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι η αποψή σας στις τροπολογίες. Ευχαριστώ, Μόλκολμ, που μου επιτρέπει να μιλήσω και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Φασανέλοβα για την επικοδομητική συνεργασία και τη συμπληρωματική υποβολή των τροπολογιών που βελτίωσε το δικό μου έργο. Η συμβατότης ε, των ε, τροπολογιών της κυρίας Ερσεναλόβα και των δικών μου ε, μπορούν να διευκρινίσουν το αρχικό κείμενο αλλά δεν μπορούσαν να περιληφθούν λόγω της εκτάσεώς τους και αυτό δείχνει την κοινή μας βούληση. Εδώ μιλάμε για ε, τα άτομα ε, τα οποία ε, πρέπει να μπορούν να προσέρχονται στην εργασία τους πιο γρήγορα παρόλο όπου έχουν πρόβλημα μετακίνησης και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό καθότι ιδίω δεν υπήρξε καμία αντίρρηση. Εδώ υπάρχουν όλα αυτά τα οποία αναφέρονται εις, ε, ε, ε, στο γενικό πλαίσιο, δηλαδή τι, τι οχήματα θα εμπλακούν, τι θα γίνει στις διάφορες περιοχές και τι θα γίνει αν κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Διότι ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρχει υπάρξει μία προστασία του ιδιωτικού τομέα και περιορισμός του κόστους σχετικά με την ε, ε, λειτουργία των ε, ηλεκτρονικών κλήσεων α, ανάγκης θα ήθελα να πω τι θα έπρεπε να περιληφθεί και τι θεωρώ περιττό. Το 1-1-2 θεωρώ ότι είναι σωστό όπως ζητάει η οίκον και να υπάρχουν και διάφορα άλλα ιδιωτικά συστήματα εκτάκτους ανάγκης, ηλεκτρονικές κλήσεις δηλαδή και όλα αυτά πρέπει να εξυπηρετούν την γρήγορη κλήση για ιατρική περίθαλψη όταν υπάρξει ένα έκτακτο περιστρατικό. Δεν θα διατηρούνται στοιχεία, δεν θα υπάρχουν τα, ε, τα στοιχεία από πού προέρχεται το τηλεφώνημα, όλα αυτά δεν θα υπάρχουν, γι' αυτό και δεν χρειάζονται τροπολογίες επ' αυτού. Θα είναι κάτι, ε, κάτι αυτόματο το οποίο θα γίνεται βάσει των αισθητήρων που υπάρχουν σε αυτοκίνητο σε περίπτωση συγκρούσεως και ε, τα συστήματα θα είναι ενιαία μετά θα μπορεί να υπάρχει και μία προσωπική επαφή με ομιλία οπότε έρχονται οι σωστικές υπηρεσίες. Για μένα αυτή δεν είναι μία αυτεπάγγελτη λύση ε, και γι' αυτό θα πρέπει να είναι και δωρεάν. Θα υπάρξουν βέβαια και δωρεάν συστήματα τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν αν υπάρχει κλίση για επίγουσα ιατρική περίθαλψη αλλά μπορεί να περιλαμβάνονται εκεί και στοιχεία μελών των, ε, ε, των αυτοκινητιστικών ε, λεσχών και τα και βεβαίως αυτά τα συστήματα θα είναι επιπληρωμή ενώ το 112 θα είναι δωρεάν. Τα συστήματα μπορούν να συνεπάρχουν του παραλίου με το 112 και το λογισμικό θα αποφασίζει στο μαύρο κουτί εάν θα επιλεγεί το 112 ή αν κάποιος το έχει αποφασίσει θα, κάνει, θα υπάρξει μία ιδιωτική ηλεκτρονική κλίση Δηλαδή μία κλίση θα γίνεται και το μαύρο κουτί ε, θα αποφασίζει οπότε θα είναι πιο εύκολα να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Ε, γι' αυτό 10% των τροπολογιών αναφέρονται σε αυτό το θέμα διότι ο καθένας ερμηνεύει διαφορετικά την έννοια αυτή. Ορισμένοι λέγουν ότι δεν πρέπει να είναι ανοιχτό σύστημα για προστασία δεδομένων, οι άλλοι μιλάνε ε, για ε, μία ουδέτερη τεχνολογικά πλατφόρμα και τέλος ορισμένοι λέγουν ότι πρέπει να υπάρχει τεχνική ουδετερότης και είναι περίπλοκο να βρεθεί μία κοινή θέση, αλλά αυτό είναι το πιο δύσκολο θέμα. Τα υπόλοιπα αναφέρονται εις ε, την ενημέρωση των πολιτών και των χρηστών και κατά την χρησιμοποίηση και την λειτουργία του συστήματος αυτών θα χρειαστούν πληροφορίες οι οποίες ε, θα περιληφθούν κατά την κατάρτιση, αλλά αυτό συμβαίνει πάντοτε όταν έχει κανείς να κάνει με μέσα δημόσιας επικοινωνίας, γι' αυτό και οι τροπολογίες αυτού νομίζω ότι ήταν θετικές. Επίσης, ε, πώς μπορεί κανείς ε, να αποκλείσει ή να εγκαταλείψει το σύστημα αυτό. Είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να κάνει συνειδητά. Αλλά αν ε, υπάρχει άμεση έκκληση σε περίπτωση συγκρούσεως, νομίζω ότι τότε είναι πιο σημαντικό να υπάρξει επέμβαση και ε, από ότι να προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα. Άρα εγώ είμαι ενάντια στον αποκλεισμό του συστήματος. Υπάρχει μία διάταξη η οποία πιστεύω θα πρέπει να είναι ενιαία ε, εφαρμόσιμη. Όσον αφορά την ε, την ε, ε, ερώτηση του πόσο μπορεί κανείς να ε, κάνει αυτές τις κλήσεις είναι ένα θέμα που θα πρέπει να ρυθμίσουμε ιδίω σε διασυνοριακές συνομιλίες και εδώ θα πρέπει να εμπλακεί η επικουρικότητα διότι τα κράτη-μέλη οργανώνουν την οδική βοήθεια διαφορετικά. Άλλοι εξαρτούν από την ε, δημόσια, από τις δημόσιες αρχές, άλλοι από τις περιφερειακές και θα πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις που να ισχύουν για όλους προστασία δεδομένων, ιδίως όταν υπάρχουν ιδιωτικά ε, ηλεκτρονικές εκκλήσεις, αυτές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένες με άλλες υπηρεσίες και να μπορεί ο καταναλωτής ε, να γνωρίζει ποιος μπορεί να παρακολουθήσει ε, αυτές τις κλήσεις, πόσο καιρό θα αποθηκευτούν, αλλά εφόσον πρόκειται για δημόσια δημόσιες ε, έκτακτες κλήσεις ανάγκης τότε δεν ε, έχουν σημασία όλα αυτά τα στοιχεία. Όσον αφορά την πρόσβαση και ιδίως για άτομα τα οποία έχουν ε, κινητικούς περιορισμούς θα πρέπει και αυτά να ληφθούν υπόψη και να ρυθμιστούν. Ζητήθηκαν νέες μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα αλλά νομίζω ότι αυτό έχει καλυφθεί και πιστεύω ότι δεν χρειαζόμαστε νέες μελέτες αποτελεσματικότητας ή μελέτες ε, για ε, κατάχρηση και λανθασμένη ε, κλίση και της βοηθείας. Δεν νομίζω ότι αυτό χρειάζεται για να θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη η κλίση με ένα συγκεκριμένο όχημα και ο δικός του του οχήματος θα μπορεί να τιμωρηθεί σε περίπτωση που υπάρχει κατάχρηση του συστήματος. Άρα ε, ε, υπό αυτές τις προϋποθέσεις δεν θα υπάρχουν καταχρήσεις και ε, θα μπορεί να υπάρξει μία ποινική διαδικασία η οποία θα τιμωρεί αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται και παρανοούν το σύστημα. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί πρέπει να υπάρξει κάποια περαιτέρω διευκρίνηση αλλά η κυρία Γιάλα Σέντερ και άλλοι είπαν ότι δεν πρέπει να ισχύσει μόνο για τα ιδιωτικά οχήματα αλλά και για τα φορτηγά και μου, λέγουν, ε, μου λέει η κυρία Γιάλα Σέντερ και για τα ποδήλατα και για τους πεζούς θα ας μου το εξηγήσει ή ε, για τα ε, οχήματα που χρησιμοποιούνται επί μακρό χρόνο ή άλλοι λέγουν ότι πρέπει να υπάρχει σε όλα τα νέα αυτοκίνητα νομίζω ότι καλό θα ήταν να περιοριστούμε στο πλαίσιο το οποίο έχουμε καταρτήσει και να μην επεκτείνουμε ατερμόνως τη χρήση αυτή. Επίσης ε, όλοι έχουν δεσμευτεί να καλούν το 112 και το ηλεκτρονικό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Ξέρω ότι ορισμένα κράτη δεν έχουν συμμορφωθεί ε, και εγώ θα ήθελα να πω ποιες είναι οι τρεις χώρες που δεν έχουν συμμορφωθεί. Ε, πιστεύω ορισμένοι ε, συνάδελφοι αντίδρασαν στο να ονομάσουμε αυτές τις τρεις χώρες αλλά ίσως είναι ε, χώρες οι οποίες δεν θέλουν να συμμετάσχουν. Και τέλος, τι τι πρέπει ε, να προβλέψουμε. Καταρχήν να υπάρχει μία αλυσίδα προστασίας στα κράτη μέλας. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο θα λειτουργεί σωστά σε όλα τα κράτη μέλη. Ε, διότι αν υπάρχουν πρώτα τεχνικά προβλήματα θα πρέπει να επιληθούν και μετά να επεκταθεί το σύστημα. Ξέρω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν εκ του παραλίλου τέλος όσον αφορά την αδειοδότηση και τελικά την εφαρμογή όποιος έχει κάνει αυτές τις τροπολογίες τον παρακαλώ να μου πει πώς το φαντάζεται γιατί οι μεν μιλούν για βαθμιαία εφαρμογή στα οχήματα και οι άλλοι μιλούν με τον ίδιο τρόπο για μία βαθμιαία εισαγωγή στα κράτη-μέλη. Οπότε θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να πούμε ότι μέχρι το τέλος του 2015 στα ε, νέα ε, οχήματα θα έχει ενσωματωθεί η λύση αυτή και ε, θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να έχουν αποφασίσει πώς θα λαμβάνουν και πώς θα προωθούν αυτές τις κλήσεις εκτάκτου ανάγκης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, πλήρη εισαγωγή. Τώρα κυρία Σεμελόβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο συνεισηγητής. Τον ευχαριστώ για όλα τα σχόλιά του. Και ακόμη και αν ε, καθόμαστε σε αντίθετα σημεία της αίθουσας, αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλίνουν και οι απόψεις μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις τροπολογίες ε, που μας στείλατε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένες, ε, κυρίως σε αυτές που εστάλησαν από τους σκιώδεις και από τους συναδέλφους αλλά θα συνεχίσουμε από κοινού να εργαζόμαστε για το τελικό αποτέλεσμα και θα συναντηθούμε και με τους σκιώδεις εισηγητές για να συζητήσουμε συμβιβαστικές λύσεις. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι το e η λεκλήση θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι ένα εθελοντικό σύστημα δεν λειτουργεί. υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και οι χρήστες ε, δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν το σύστημα για να σώσουν ζωές. Όμως ε, δεν συμφωνούμε σχετικά με το πότε θα πρέπει να εισαχθεί το σύστημα. Ο κύριος Χάρμπορ και η κυρία Παρβάνοβα, παραδείγματος χάρη, στις τροπολογίες 31 και 32 αναφέρονται στην αναγκαιότητα εισαγωγής του e μετά ε, την ε, υλοποίηση της υποδομής ε, και θα ήθελα να αναφερθώ στη σύσταση του περασμένου Σεπτεμβρίου της Κομισιόν όπου τα κράτη-μέλη μαζί με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την υποδομή και ακόμη και αν δεν απάντησαν όλα τα κράτη-μέλη σε αυτές τις ερωτήσεις και το αναφέρουμε αυτό σε μία από τις τροπολογίες από τα 18 κράτη-μέλη μόνο ένα είπε ότι δεν έχουν κέντρο λήψης κλίσεων έκτακτης ανάγκης PSAP. Κανένας παροχός κινητής τηλεφωνίας δεν αρνήθηκε να εφαρμόσει την ε, σημαία ε, η call που είναι απαραίτητη για τη, απαραίτητη για τη διαβίβαση των δεδομένων. Έτσι λοιπόν υπάρχει ετοιμότητα να αυτή το e-call και ίσως ε, οι εκπρόσωποι της Κομισιόν θα μπορούσαν να μας πούν κάποια παραπάνω στοιχεία, να μας δώσουν κάποια παραπάνω στοιχεία για το feedback και για την έρευνα. Κάποια ε, στροπολογίες αφορούν το κόστος ε, εξοπλισμού στα κέντρα λήψης κλήσεων εκτεκτης ανάγκης και δεν θέλω να αναφέρω τα πιλωτικά προγράμματα. Αυτά αναφέρονται και στην έκθεση. Υπάρχουν τρεις ε, πιθανές λύσεις για τα κέντρα λήψεων, πώς να οργανωθούν δηλαδή και να λαμβάνουν κλήσεις εκτεκτης ανάγκης τα, οι δοκιμές μας δείχνουν ότι για να υπάρχει πλήρης λειτουργικότητα μπορούμε να έχουμε μόνο τα δύο, ένα ή δύο τέτοια κέντρα που θα παραλαμβάνουν τις κλήσεις, θα δέχονται τις κλήσεις και κατόπιν θα διανέμουν τις κλήσεις αυτές σε όλο το δίκτυο. Και το κόστος των κλήσεων είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και δεν υπάρχει απέτηση για κάλυψη με προσωπικό. Υπάρχει μόνο κάτι τέτοιο που αναφέρεται ε, στην τροπολογία 85 και μιλάμε για πρόσθετη κατάρτιση του προσωπικού. Συμφωνώ επίση με την τροπολογία τη κυρία Τούν ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να βελτιώσουν τη λειτουργία τη γραμμή 112, τροπολογία 52. Ανέφερα και το πιλωτικό πρόγραμμα εδώ και θα ήθελα να σας εξηγήσω τι είναι. Πρόκειται για ένα τεστ, ε, όχι για ένα project επίδειξης ε, που ανέφερε ο κύριος Χάρμπορ ε, στην τροπολογία 27. Συμφωνώ με την κυρία Παρβάνοβα στην τροπολογία 99 ότι πρέπει να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές ακόμη και διασυνοριακά σε ό,τι αφορά τα κέντρα έλλειψης κλήσεων εκτά της ανάγκης. Η τροπολογία που αφορά τη τεχνολογική ουδετερότητα τροπολογία 43, τροπολογία 45, Παρβάνοβα και Χάρμπορ. Ο στόχος της εκθεσής μας είναι να εισαγαγούμε το e-call ως ένα εργαλείο ασφαλείας και προκειμένου να το κάνουμε αυτό, πρέπει να διατηρήσουμε ελάχιστα κοινά πρότυπα προκειμένου να είναι διαλειτουργικά τα συστήματα σε όλη την Ευρώπη. Και πιστεύω λοιπόν ότι θα καταλήξουμε σε μια καλή συμβιβαστική λύση που θα προσφέρει όσο δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια στον τελικό χρήστη. Το τελευταίο θέμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι η ανοιχτή πλατφόρμα για το e-call που θα επιτρέψει να προσθεθούν και άλλες υπηρεσίες. Νομίζω ότι πρέπει να επιτρέψουμε στους καταναλωτές να μπορούν να επιλέγουν αυτές τις υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και φυσικά ανυπομονώ να γίνει η συζήτηση και ανυπομονώ να εργαστούμε περαιτέρω επί των τροπολογιών. Πιστεύω ότι είναι προς το δικό μας συμφέρον να έχουμε μια καλά ισορροπημένη έκθεση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την ιδανική ευκαιρία εδώ να επεκτείνει τη μέγιστη υποστήριξή του σε αυτό το πολύ χρήσιμο σύστημα και πιστεύω ότι θα δράξουμε αυτή την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Σενάλοβα και να ευχαριστήσω και τους δύο συγγητές. Ας δούμε τώρα τι έχουν να πούν οι σκιώδεις συγγητές. Είναι όλοι όμως εδώ, αυτό θέλω να ελέγξω πρώτα. Και μπορείτε στη συνέχεια και οι υπόλοιποι να πάρετε το λόγο και να μου το πείτε. Η σκιώδης είναι η κυρία Τούν Χονστάιν από την ΙΜΚΟ από την Άλντε ο κύριος Μπένιον από την Επιτροπή Μεταφορών, η κυρία Ρούλερ και ο κύριος Τέιλορ είναι και οι δύο παρόντες. Ο κύριος Τέιλορ νομίζω θα πάρει πρώτο το λόγο, σωστά. Και η κυρία Φώστερ για το ECR στη συνέχεια. Και θα ακούσουμε και άλλους ομιλητές. Στη συνέχεια η κυρία Γκέπχαρτ θέλει να πάρει το λόγο. Υπάρχει κάποιος άλλος που δεν είναι σκιώδης και θέλει να μιλήσει. Θα πάρω και εγώ το λόγο στη συνέχεια αλλά πρώτα θα μιλήσει για το ECR η κυρία Φώστερ. Ας ακούσουμε πρώτα την κυρία Τούν Χόνεσταϊν. Ευχαριστώ πολύ και να σας ευχαριστήσω για όλη την εργασία καθώς επίσης και την μακροχρόνια εμπλοκή σας σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και πραγματικά ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση αυτή, όπως ε, άλλωστε επιθυμεί ο κύριος Κόχ τα τελευταία δέκα χρόνια. Ελπίζω ότι θα έχουμε έμπρακτα αποτελέσματα στα χέρια μας σύντομα. Και γι' αυτό το λόγο περιμένω και εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουμε μια νομοθετική πρόταση. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα μια νομοθετική πρόταση για το ζήτημα αυτό. Μια νομοθετική πρόταση δεσμευτική για όλα τα κράτη-μέλη. Όπω είπε η κυρία Σενάλοβα, είναι πολύ καλό το ότι υπάρχει τουλάχιστον μια πολιτική βούληση εκ μέρου των κρατών μελών για να συνεργαστούν, ε. αλλά λυπούμε από αυτό το μνημόνιο συνεννόηση δεν υπεγράφει από όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει πάντως μια γενικότερη πολιτική βούληση, υπάρχει μια ετοιμότητα, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο σαφή και ξεκάθαρα όσο θα επιθυμούσαμε. Έχουμε ένα πρόβλημα με την υπαριθμόν 112 τροπολογία. Τα όσα λέγονται εκεί πέρα δεν λειτουργούν στην πράξη και συμφωνώ με αυτά που είπαν οι εισηγητές. Έχω καταθέσει λοιπόν μια επιπλέον τροπολογία και θεωρώ ότι θα πρέπει να ασκηθεί πίεση στα κράτη-μέλη προκειμένου ο αριθμός 112, ο αριθμός κλίση 112 να λειτουργεί στην πράξη. Θα πρέπει επίσης ο σχετικός εξοπλισμός να εγκατασταθεί στα οχήματα, αλλά πρώτα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα όσα θα πρέπει να υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο για τη δημόσια ασφάλεια και στη συνέχεια να έρθει το e-call, η ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία κλήσεων, να συμπληρώσει το σύστημα αυτό. Και η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να είναι δημόσια και θα πρέπει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και να είναι προσβάσιμη σε όλους. Η συσκευή αυτή συμφωνώ ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί στα οχήματα. Συμφωνώ πλήρως με τους συγητές. Θα πρέπει να ενσωματωθεί σε κάθε όχημα αυτή η συσκευή. Ουσιαστικά Αυτές είναι οι βασικές μου παρατηρήσεις. Βλέπω ότι στα περισσότερα σημεία συμφωνούμε, εκτός από αυτά τα ελάχιστα τα οποία μόλις τώρα ανέφερα και να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι χρειαζόμαστε μία νομοθετική πρόταση για το ζήτημα αυτό και ελπίζω αυτό να γίνει πραγματικότητα σε όλα τα κράτη-μέλη σύντομα. Ευχαριστώ. Uh, ε, Mr. next. Yes, uh, ναι. Ο κύριος Μπένιον, ναι, ναι εγώ από τη συνάδελφο, την κυρία Περβάνα, που δεν μπορεί να είναι εδώ. Έχω λοιπόν ένα συνδυασμό σχολείων που προέρχονται και από δυο μα. Ορισμένα συνάδουν μεταξύ τους, αλλά όχι. Θέλω να ευχαριστήσω ε, τον εισηγητή, την εισηγητρία μάλλον που έλαβε υπόψη πολλά θέματα που θέσαμε και το θέμα των ψεύτικων συναγερμών, ε, των ψευδών συναγερμών, ε, συναδημόσα είπαμε, αλλά μου άρεσε η τροπολογία του κύριου Τάιλερ. Νομίζω ότι εξακολουθεί να πρέπει να υπάρχει στο κείμενο αυτό παρά απλώ να θεωρούμε ότι πρόκειται για κάτι δεδομένο. Νομίζω ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο ρητά. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιο συνδεσμό, αλλά νομίζω ότι το κείμενο του κ. Τάιλερ είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή σε ό,τι αφορά αυτούς τους ε, σε συναγερμού και την ανάγκη να διαφοροποιήσουμε ε, μεταξύ των ε, ατυχημάτων και περιστατικών που πρέπει να καλούνται οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Και θα ήθελα να συνεχίσει να περιλαμβάνεται λοιπόν κάτι τέτοιο. Βέβαια, εξακολουθώ να είμαι ότι θα πρέπει όλη η αλυσίδα διάσωση να υπάρχει και να λειτουργεί πριν να ξεκινήσει το σύστημα, να λειτουργεί. Γιατί αν λειτουργεί μόνο εν μέρη, αν λειτουργεί σε ορισμένε περιοχέ και όχι σε κάποιε άλλε, ε, τότε θα υποσκάψει το όλο σύστημα. Γιατί θα πιστεύουν ε, οι άνθρωποι ότι θα καταφτάσουν οι υπηρεσίε εκτακτή ανάγκη, ενώ δεν θα έχουν κληθεί γιατί δεν θα λειτουργεί το σύστημα. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη πρόσβαση, την ανοιχτή πρόσβαση. Νομίζω ότι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο ιδιωτικό τομέα να μπορεί να χρησιμοποιεί συστήματα ανοιχτή πρόσβαση για τι πρόσθετε υπηρεσίε, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να καλύπτεται από τη δημόσια υπηρεσία. Η πλατφόρμα του e νομίζω ότι πρέπει βασικά να σχεδιαστεί για να παράγει μόνο τα ελάχιστα δεδομένα. Γιατί αν ε, αρχίζουμε να προσθέτουμε διάφορα στοιχεία στη δημόσια υπηρεσία, τότε όχι μόνο απειλούμε την ασφάλεια των δεδομένων, αλλά θα αυξήσουμε και το κόστος. Και ένα από τα κύρια προβλήματα με το e είναι το κόστος. Ε, που μπορεί να επιφέρει σε ένα όχημα χαμηλή αξία. Έτσι λοιπόν, ό,τι και να κάνουμε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα είναι βασικό και απλό και έχει σχεδιαστεί μόνο για να καλύψει τις ε, έκτακτες ε, ε, περιστάσεις και όχι να έχουμε μία σειρά πρόσθετων λειτουργιών. Η κυρία Περβενοβά δεν ε, έχει δει ακόμα μία πλήρη μελέτη για τα θύματα, για τη μείωση των θυμάτων. Δεν ε, έχει δει μία κατάλληλη μελέτη επιπτώσεων. Θα θέλαμε να υλοποιηθεί μια τέτοια μελέτη επιπτώσεων. με τετοια μελετη ότι διαφωνείτε και το έχετε καταστήσει σαφές. Τέλος. Για την επέκταση αυτού του συστήματος σε όλα τα ίδια οχημάτων, η κυρία Παρβάνοβα είναι υπέρ το να εξετάσουμε και τις μοτοσυκλέτες. Εγώ θα ανησυχούσα στο να προσθέσουμε αυτό το σύστημα στις μοτοσυκλέτες χωρίς ε, να έχουμε την κατάλληλη διαβούλευση και τη μελέτη αντικτύπου. Κυρίως πρέπει να ρωτήσουμε τους ίδιους τους μοτοσυκλετιστές. Δηλαδή να έχουμε μια τροπολογία χωρίς να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες δεν νομίζω ότι είναι σωστή οδός να ακολουθήσουμε και δεν είμαι και τόσο κατά στο να επεκταθεί σε κάποια ελαφρά εμπορικά οκήματα. Νομίζω ότι ίσω θα μπορούσαν να καλυφθούν αυτά τα ελαφρά οχήματα. Δεν είμαι βέβαια σίγουρο. Όχι στα τρακτέρ βέβαια, όχι στου ελκυστήρε. Γιατί πολύ συχνά διαφέρει η φύση ε, της μετακίνησης με τα τρακτέρ και επειδή έχουμε πολλές δύσκολες μεταφορές ε, με τα τρακτέρ, θα είχαμε πάρα πολλούς, ε, ψε, πολλούς ψευδείς ε, συναγερμούς. Νομίζω ότι τα κάλυψα όλα. Ευχαριστώ. Δεν πρόσεξα να αναφερθήκατε σε τροπολογίες. Θα περιμένουμε να δούμε. Κύριος Τέιλορ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τους δύο συγητές για την πολύ χρήσιμη και έγκαιρη και θετική έκθεση. Αν δούμε τα κυρία σημεία, θα συμφωνούσα με την έννοια του συστήματος ε, ηλεκλήσης και συμφωνώ ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα. Πιστεύω ότι το σύστημα e-call μπορεί να αποδειχθεί ένα σημαντικό στοιχείο στο να βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους της Κομισιόν, να μειώσουμε τα θανατηφόρα ατυχήματα ε, και τους σοβαρούς τραυματισμούς. Ε, το e θα μπορέσει να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσουμε τα ατυχήματα. Νομίζω ότι η κλίση του e δεν πρέπει να καλυπτεί μόνο τα οχήματα ε, των οδηγών, αλλά αφορά όλους τους χρήστες ε, των ε, δρόμων, του δικοδικτύου και πρέπει να δούμε και αν θα έχουμε ένα σύστημα e-call και σε όσους κινούνται με δίκυκλα, γιατί και αυτοί μπορεί να φυγούν από ατυχήματα και η οδήγηση είναι ευθύνη, δεν είναι δικαίωμα. Ε, των ανθρώπων να οδηγούν όπου και όποτε θέλουν ε, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη, να λαμβάνουν καμία ευθύνη και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, ένα σημαντικό μήνυμα που πρέπει να διαβιβάσουμε και είναι τμήμα τη κοινή μας ε, ευθύνης. Και θα ήθελα να πιστεύω ότι τα επόμενα έτη θα σκεφτόμαστε την εποχή πριν το e πριν να ήταν διαθέσιμο αυτό το μέσο ε, στους ε, χρήστες των οδών, έτσι ε, όπως σκεφτόμαστε σήμερα για τις ζώνες ασφαλείας στα αυτοκίνητα. Και αν το σκεφτείτε, ακριβώς περί του δύο μέτρου πρόκειται. Δηλαδή πρόκειται για έναν τρόπο να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή όταν χρησιμοποιούμε τα συστήματα μεταφορών. Έτσι λοιπόν, εγώ θα ήμουν ε, υπέρ ε, του να έχουμε καλά οχήματα, να επεκτείνουμε το ΕΚΟΛ και σε άλλα οχήματα, ίσως όχι για τους πεζούς, να μην καλύψουμε τους πεζούς, αλλά όταν μιλάμε για οποιοδήποτε όχημα με κινητήρα, νομίζω ότι αν υπήρχε ένα σύστημα σε αυτό, τότε θα ήταν προς όφελός του. Σε σχέση με τις ε, τροπολογίες που προσθέσαμε από την Επιτροπή Μεταφορών, Πιστεύουμε ότι το e θα πρέπει να ενσωματωθεί στι εφιστάμενες υπηρεσίες 112 και θα πρέπει να ενισχυθούν οι υπηρεσίες αυτές αν δεν καλύπτουν το στόχο του. Στην παράγραφο 4 και ευχαριστώ τον ε, κύριο Μπένιον για την υποστήριξή του σε αυτό πρέπει να αξιολογήσουμε ε, τους ε, πιθανούς ψεύτικους συνεγερμούς και να δούμε πώς ε, θα διαφοροποιήσουμε τα σοβαρά τυχήματα από τις μικροσυγκρούσεις. Και τέλος, νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά που συνεχίζουν να μένουν αναπάντητα είναι το εξή. Τροπολογία μας για την παράγραφο 5 προτείνει στην Κομισιόν ε, να παρουσιάσει μια ποσοτική εκτίμηση του κόστου της επιδομής και πώς θα καλυφθεί το κόστος αυτό. Και γιατί αυτό είναι κάτι που έχει συνέπειες και πρέπει να διερευνηθεί. Γενικά πάντως πιστεύω ότι είναι καλή η ιδέα αυτή. Ας κάνουμε μια θετική προσπάθεια να υιοθετηθεί αυτός ο μηχανισμός στο σύστημα. Ευχαριστώ κύριε Τέιλορ και κυρία Φώστερ. Ε, Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Η Άννα Ρόσπαχ είναι η η συγγητριά μας, αλλά συνάδουν ουσιαστικά οι απόψει μα, Να ευχαριστήσω του συγγητές για την τεράστια εργασία που έχουν κάνει για τη σημερινή έκθεση και βέβαια χρειάστηκε να εξετάσουν και όλε αυτέ τις τροπολογίε. Αναμφίβολα, όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ πέρα θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι σε περίπτωση αυτοκινηστικών ατυχημάτων πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιδρούμε γρήγορα και να σώζουμε ζωές. Αυτό νομίζω ότι μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο επίπεδο αυτοβελτίωσης της κατάστασης σε σχέση με το πώς έχει σήμερα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την αριθμό κλήσης 112 και είναι πολύ σημαντικό οπουδήποτε και αν βρίσκεται κανείς στη χώρα του στο εξωτερικό να μπορεί να χρησιμοποιεί τον αριθμό αυτό. Εξετάζοντας όμως περισσότερο την κατάσταση αυτή, και δεν μα έχει βοηθήσει ιδιαίτερα και σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδαμε ότι υπάρχουν περισσότερα ερωτήματα από ό,τι απαντήσει. Ακούγοντα κανεί συζήτηση αυτή, βλέπει ότι η υποδομή καν δεν υφίσταται. Υφίστανται ακόμα πολλά ερωτήματα για το αν αναφερόμαστε για παράδειγμα σε υγειονομικέ υπηρεσίε. Σε ορισμένε χώρε δεν θα υπήρχε πρόβλημα να εμφανιστεί ένα ασθενοφόρο και να βοηθήσει τον ε, τραυματία. Σε άλλες χώρες όμως υφίσταται διαφορετικά συστήματα. Μπορεί να έρθει ένα στενοφόρο, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο τραυματίας να πληρώσει για την υπηρεσία αυτή. Δεν προσφέρεται δηλαδή άμεσα και δωρεάν. Σίγουρα δεν υπάρχει λοιπόν εναρμονισμένο σύστημα. Δεν λέω ότι θα πρέπει σώνει και καλά να εναρμονιστεί το σύστημα, απλώ υπάρχουν κάποιε λεπτομέρειε οι οποίε πρέπει να διευθετήσουμε προκειμένου το νέο αυτό σύστημα να μπορεί να λειτουργεί ομαλά, χωρί προσκόμματα. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο εξετάσαμε είναι αν θα συμβάλλει και ο δημόσιος τομέας ή αν θα πρέπει να υπάρχει και μια συμβολή του ιδιωτικού τομέα, ιδίω όσον αφορά την ε, τεχνολογία. Επίσης κάποιες υπηρεσίες μπορούν να δωρεάν, άλλε πάλι όχι. Αυτό που με μπερδεύει είναι το εξή. Αν κάτι δεν λειτουργήσει τι θα γίνει. Ή, αν για παράδειγμα έχουμε ένα ατύχημα, αν κάποιο έχει χάσει τι αισθήσει του, τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή. Αν πρέπει σών και καλά να υπάρχει μια ανταπόκριση, μια συνομιλία. Αν θέλουμε πραγματικά ένα τόσο γενικό ευρύ εφαρμοσμένο σύστημα, θα ήθελα να γνωρίζω ακριβώ πώ θα λειτουργήσει, τι θα γίνει σε περίπτωση σύγκριση. Κανεί δεν μου έχει εξηγήσει ακριβώ από τεχνική πλευρά πώ πρόκειται να λειτουργήσει το σύστημα. Πρέπει να επιμείνουμε λοιπόν ιδιαίτερα στα τεχνικά ζητήματα της υποδομής. Δεδομένα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε, το συζητήσαμε την προηγούμενη φορά, δεν είναι μόνο η ασφάλεια των δεδομένων, είναι ποιο θα έχει στην διάθεσή του τα δεδομένα αυτά και πόσα δεδομένα τελικά θα πρέπει να διοχετευθούν. Δεν έχει δοθεί απάντηση γι' αυτό ακόμα. Στην προηγούμενη συζήτηση μιλήσαμε και για την ε, δυνατότητα να επενεργοποιήσει κανείς το σύστημα αυτό μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Νομίζω το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι εθελούσιο. Το 2015 είναι μια πολύ κοντινή καταλεκτική ημερομηνία. Κανείς δεν αναφέρθηκε στην κατασκευαστική βιομηχανία, στην αυτοκινητοβιομηχανία. Στην προηγούμενη συζήτηση είχαμε πει πολύ απλά ότι με 30 ευρώ θα μπορέσουν να εγκαταστήσουν την συσκευή αυτή στα αυτοκίνητα. Μα δεν είναι 30 ευρώ το κόστος, είναι 300 ευρώ και στο μέλλον, καθότι θα παραχθούν όλο και περισσότερα τέτοια μικροτσίπ, μπορεί το κόστο όντω να κατέβει στα 30 ευρώ, αλλά μπορεί να υπάρχουν και κάποιε επιπλέον δαπάνε που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Πιστεύω λοιπόν το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι εθελούσιο και θα πρέπει να εξεταστεί και το ζήτημα του κόστους. Σε ορισμένους αυτό μπορεί να αρέσει, σε άλλους πάλι όχι. Είναι πάντως ένας καθοριστικός παράγοντας στην όλη συζήτηση. Κανείς δεν αναφέρθηκε στον τομέα αυτοκατασκευών, στην αυτοκινητοβιομηχανία. Έχω μιλήσει με κατασκευαστές από τη δική μου εκλογική περιφέρεια Και νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα, ιδίω με τα αυτοκίνητα αυτά τα οποία έχουν χαμηλή τιμή, τα πιο φτηνά αυτοκίνητα, τα οποία θα πρέπει να εξοπλιστούν με το σύστημα αυτό. Σίγουρα η όλη ιδέα, η όλη πρόταση είναι πολύ καλή. Σαφώ θέλω να χρησιμοποιηθεί το σύστημα αυτό. Απλώ θα ήθελα να μου δοθούν κάποιε πιο συγκεκριμένε απαντήσει στα ερωτήματα αυτά τα οποία κατέθεσα. Με τον κύριο Χάρμπορ προσπαθήσαμε να δούμε πώ θα λειτουργήσει το σύστημα, αν θα είναι όντω διαλειτουργικό και αν όντως πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια κάποια τεχνολογία, αυτή θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε όλες τις χώρες. Δεν είμαι κατά του συστήματος, που πανλαμβάνω. Πρέπει να εξετάσουμε απλώς όλες τις πλευρές και τις τεχνικές πλευρές. Από θεωρητικής πλευράς τα πράγματα ακούγονται ρόδινα και πολύ ωραία. Στην πράξη όμως βλέπει κανείς ότι γίνονται πολύ πολύπλοκα. Υπάρχουν πολύπλοκα τεχνολογικά συστήματα τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν ομαλά σε όλες τις χώρες. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχει καν η βασική υποδομή. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν είναι ρεαλιστικό να, να προχωρούμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε αυτή τη στιγμή την εφαρμογή του συστήματος τη στιγμή που λείπει μια πολύ βασική υποδομή. Και ολοκληρώντας σε σχέση με κάτι που είπε και ένα συνάδελφος, τρεις χώρες δεν έχουν συμφωνήσει. Μα δεν είμαστε στη Σοβιετική Ένωση. Νομίζω ότι να πρόκειται στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν αν θέλουν να συμμετάσχουν στο σύστημα αυτό ή όχι. Δεν υποχρεούνται Ούτε πρέπει να κατανομάσουμε αναγκαστικά τα κράτη αυτά. Έχουν το δικαίωμα να πούνε ότι δεν θέλουν να συμμετέχουν, όπω υπάρχουν και κάποιε άλλε χώρε οι οποίε είπαν εξ αρχή ότι θέλουν να συμμετέχουν. Ενδεχομένω οι χώρε αυτέ να μην έχουν ε, συμφωνήσει ακόμα με το σύστημα αυτό, να μην θέλουν να συμμετάσχουν και δεν του έχουν δοθεί όλε αυτέ οι απαραίτητε απαντήσει. Ευχαριστώ. Uh, now we then turn... Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Να, από τους σκιώδεις τώρα να περάσουμε στου υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Η κυρία Γκέπαρτ, ε, καταρχήν ε, να ξεκινήσουμε από εσά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να ξαναγυρίσουμε στο σημείο κινήσεως και να σκεφτούμε γιατί συζητάμε τώρα. Γιατί αυτή είναι η εντύπωση την οποία αναπεκόμισα από τη συζήτηση την οποία κάναμε. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά ατυχήματα και στα πολλά ατυχήματα υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία τραυματίζονται ελαφρά ή πολύ βαρύτερα και χρειάζεται να τα βοηθήσουμε αμέσως. Αυτό είναι το σημείο κινήσεως της συζήτησης και με τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες τις οποίες έχουμε μπορεί κανείς να έχει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Οπότε να μπορεί κανείς να πει υπάρχει ένα ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο και μπορείτε αναλόγως να αντιδράσετε. Αυτό είναι το σημείο κινήσεώ μας. Είπαμε λοιπόν αφού διαπιστώσαμε ότι τα κράτη-μέλη δεν προχωρούν τόσο γρήγορα ότι εδώ είναι ανάγκη να προχωρήσουμε σε μία νομοθεσία και νομίζω ότι σωστό είναι να υπάρξει ευρωπαϊκή νομοθεσία διότι όλο και περισσότεροι κάνουν διακοπές κάπου κάπου ή δουλεύουν κάπου αλλού και δεν ξέρουν που θα έχουν ένα ατύχημα και ακόμη και αν είναι κανείς τραυματισμένος και έχει ένα κινητό στο χέρι ποιον θα, σε ποιον θα τηλεφωνήσει ή αν είναι ανέστητος τι θα γίνει δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα κράτος μέλος όπου ε, υπάρχει ένα νοσοκομιακό το το οποίο έρχεται και που έχει στο χέρι του ένα κινητό και θα τον πάρει αν δεν εξασφαλίσει ποιος θα πληρώσει τα έξοδα. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι τελείως αντίθετο προς τις αξίες Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά και ελπίζω να μην είμαι τόσο αφελής και να παρουσιάζομαι ε, έτσι έναντι του εισηγητή. Απλούστατα υπάρχουν συστήματα, έρχεται το μήνυμα και λέγει υπάρχει ένα τραυματισμός χωρίς προσωπικά στοιχεία. Ένα αυτοκίνητο έχει, έχει ένα ατύχημα, υπάρχουν τραυματισμοί και πρέπει να ασχοληθούμε και να επέμβουμε και ενδεχομένως να φτάσουμε εκεί το ταχύτερο δυνατόν. Αυτό είναι το μέλημά μας. Παρακαλώ λοιπόν να σκεφτούμε και να δούμε πώς μπορούμε να ε, καταρτήσουμε ένα τέτοιο σύστημα με αισθητήρε, οι οποίοι σε περίπτωση ανάγκης θα εκλείονται και θα ξεκινούν και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ελέγξουν οι ειδικοί για το πώς μπορούν να δημιουργηθούν και έτσι θα υπάρξει ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργήσει γρήγορα, αποτελεσματικά και απλά. Και Υπάρχουν διαφορετικά σήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί και πρέπει να δούμε αν θα είναι συμβατά. Εάν τα σήματα αυτά θα φτάνουν στα σημεία που πρέπει να φτάσουν και αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Δεν είναι η μεγάλη μας δυσκολία σήμερα όπως ήταν πριν από 5, 10, 15, 20 χρόνια γιατί τεχνολογικά στην καθημερινή μας ζωή έχουμε προχωρήσει κάθε, ε, πάρα πολύ τεχνολογικά. Οπότε καλό θα ήταν να περιοριστούμε, να δούμε ποια είναι η απλούστερη μέθοδος την οποία μπορούμε να εκπονήσουμε ώστε να εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης να μην είναι τεχνολογικά πολύ περίπλοκα γιατί αν είναι πολύ περίπλοκα μπορούν να έχουν περισσότερες βλάβες και να μην λειτουργήσουν σωστά να μην είναι πάρα πολύ ακριβά γιατί θέλουμε να μπορούν να εισαχθούν σε όλα τα νέα αυτοκίνητα και κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό να είναι είναι υποχρεωτικό σε όλες τις νέες αδειοδοτήσεις από ένα σημείο και πέρα και αυτό το αφήνω στη διάκριση των εμπειρογνωμόνων μας να μας πούν ποια θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να εισαχθεί ένα τέτοιο σύστημα. Αλλά θα πρέπει να εκπονήσουμε ένα απλό σύστημα για να επιτύχουμε ακριβώς αυτό το οποίο είναι αναγκαίο για να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν βοήθεια για τους ανθρώπους που τη χρειάζονται. Ποιος θα εμπλακεί καταρχήν είναι τα αυτοκίνητα και καταλαβαίνω ότι έχει νόημα Δεν μου έρχεται όρος τώρα για τα ε, για ε, δίκυκλα δηλαδή μοτοσικλέτες είμαι τόσο ε, κρυωμένη ώστε χάνω τα λόγια μου λοιπόν για μοτοσικλέτες όπου υπάρχουν τόσες σοβαρές, τόσα σοβαρά τυχήματα όπου το χρειάζονται και για άλλα μηχανήματα έχω ερωτηματικά αλλά στα αυτοκίνητα στα, στις μοτοσικλέτες και σε οχήματα τα οποία ενοικιάζονται και έχουν πολλά τυχήματα ε, δεν είναι ίσως τόσο γενική ανάγκη και γιατί τον, το τονίζω, διότι όσο περισσότερα αυτοκίνητα περιλάβουν αυτό το σύστημα τόσο φθηνότερο θα είναι και είναι και ένα θέμα, θέμα κόστους το οποίο πρέπει να συνυπολογίσουμε για να δούμε πόσο θα ενσωματώσουμε και την οικονομική σκοπιμότητα ώστε άτομα τα οποία έχουν ε, ένα ατύχημα και δεν μπορούν πλέον να επικοινωνήσουν μόνοι τους ή είναι σε απόμακρη περιοχή όπου δεν περνά κανένα αυτοκίνητο, πώς θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν ότι η βοήθεια θα φτάσει γρήγορα. Η κυρία Βανιού και ο κύριος Σάβαμα. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές ε, που έβαλαν τη δυναμά τους, ε, έτσι ώστε η έκθεση αυτή που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική για τους Ευρωπαίους πολίτες ε, να μπορεί να έχει την κατάλληλη έκβαση. Κατά την πρώτη συζήτηση για το θέμα αυτό είχα πάρει το λόγο για να καταδείξω ε, την κάπως παράξενη στάση των αρχών κάποιων χωρών όπως και της δικής μου πάνω στο σύστημα e όπως προτείνεται από την Κομισιόν και πιο συγκεκριμένα για τη χρησιμοποίηση ε, του αριθμού 112 και τελικά δικαιώθηκα γιατί βρήκα κάποιες ε, τροπολογίες ε, κυρίως Γάλλων συναδέλφων που θετούσαν την γαλλική θέση και αυτό έχει να κάνει με δύο επιχειρήματα. Το e-call θα πρέπει να βασίζεται σε ιδιωτικά δίκτυα που θα αναπτύσσουν οι κατασκευαστές κάτι πολύ καλό γιατί έχουμε την όμιλο Πεζό στη Γαλλία και πολύ ωραία και κάθε ε, δημόσια ανάπτυξη όπως το 112 θα σήμαινε ότι θα πρέπει να επικερπίσουμε το κόστος του κέντρου κλήσεων. Βέβαια αυτά τα δύο επιχειρήματα μεταφράζονται σε τεχνολογική ουδετερότητα και στην προσφυγή σε ιδιωτικά κέντρα για τις ψευδείς κλήσεις ε, για να τις ε, εξελίψουμε όμως. Το θέμα είναι ότι στην Γαλλία τα κέντρα εδώ και 30 χρόνια λίγο έχουν εξελιχθεί, στο παρελθόν ήταν πολύ καλά, ε, όμως ε, δεν έχουμε πολλά διδάγματα να λάβουμε και κυρίως ε, όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που την ευχαριστώ για την πρότασή της, καθώς η πρόταση αυτή δεν είναι τέλεια βεβαίω, αλλά παρόλα αυτά οδεύει προ τη σωστή κατεύθυνση. Το Πανευρωπαϊκό Οικό λειτουργεί τεχνικά σε νέα χώρε όπου είναι σε στάδιο ε, νέας ανάπτυξης ε, βάσει σε στάνταρ TSC και CNN ε, και το σύστημα αυτό προβλέπει, επιτρέπει ήδη την συνέχιση και τη διαλειτουργικότητα της υπηρεσίας ε, μεταξύ των κρατών μελών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ψευδείς κλήσεις, το προτινόμενο πρότυπο μας επιτρέπει να διαφοροποιήσουμε μια κλασική κλίση από μια κλίση call και να ξέρουμε αν μια κλίση call έγινε αυτόματα ή ε, με το χέρι. Επίσης, η Γαλλία έχει το πιο μεγάλο ποσοστό των κλασικών ψευδών κλίσεων, ε, γιατί ξεκινάμε και με εκστρατεία τώρα. Ε, όμως, αυτό το επιχείρημα των ψεύτικων κλήσεων ε, μας δείχνει συγκεκριμένα το πόσο ανάγκη είναι να επανασχεδιάσουμε τον οργανισμό του κέντρου κλήσεων. Έχουμε περίπου 100 τέτοια κέντρα στη Γαλλία, νομίζω ότι έχουμε και εκατοντάδε στη Γερμανία και δεν θα αναφέρω όσα είπε η κυρία Γκέπαρτ, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί τη και τα κέντρα αυτά είναι κατακαιρματισμένα σε διάφορε υπηρεσίε εκτέτη ανάγκη. Είναι λοιπόν αναποτελεσματικό και δαπανηρό όλο αυτό το σύστημα και επίση ε, νομίζω ότι το να επενδύσουμε, πόσο μάλλον να επενδύσουμε στην επανεργάνωση, Φυσικά θα χρειαστούμε και κατάλληλη προθεσμία. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το τίμημα μια ε, ζωή ε, που σώζεται έχει και ένα οικονομικό κόστο, αλλά εμεί ω Ευρωπαίοι νομοθέτε έχουμε το καθήκον να δείξουμε ότι η Ευρώπη έχει ένα σύστημα αποτελεσματικό, ένα σύστημα ασφαλεία αποτελεσματικό και που να λειτουργεί και ότι μπορεί και οφείλει να προστατεύει του πολίτε τη. Εγώ νομίζω ότι ε, πρέπει να έχουμε το θάρρο να μην κρυβόμαστε πίσω από επιχειρήματα μερικά για να αιτιολογούμε κάποιες εύκολες επιλογές δηλαδή επιλογές ανεύθυνες. Σας ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τέλος ο κύριος Σαβανά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η βασική μου παρατηρήση είναι η ακόλουθη. Και ουσιαστικά πιστεύω ότι για αυτό το λόγο βρισκόμαστε όλοι εδώ, όχι απλώς για να ενώσουμε την Ευρώπη, αλλά για να την κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερη για όλους. Συμφωνώ πάντως με τις ανησυχίες της κυρίας Φώστερ μέχρι ενός βαθμού. Δηλαδή, η αξιολόγηση της εφαρμογής στην πράξη του συστήματος αυτού. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τα κέντρα κλήσεων εκτάκτου ανάγκης θα είναι όντω έτοιμα παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2015. Συμφωνώ λοιπόν με την κυρία Φώστερ ότι ε, θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα πραγματικά και εγώ να έχουμε μια ισχυρή νομοθεσία η οποία να λειτουργεί για όλους με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμβολή σας και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όχι μόνο ω σκιώδης εισηγητής αλλά και επειδή θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας και να σας υπενθυμίσω το ότι όσον αφορά την ετοιμότητα του συστήματος, από τότε που είχαμε την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών από το 2001 τα δίκαια μετά, τα κράτη-μέλη είχαν συμφωνήσει ότι για τις κλήσεις εκτάκτου ανάγκης θα δημιουργήσουν την απαραίτητη υποδομή προκειμένου να μπορούν να εντοπίσουν γεωγραφικά τις κλήσεις αυτές οι οποίες προέρχονται μέσα από ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, κλήσεις εκτάκτου ανάγκης. Ήταν πολύ δύσκολο έκτοτε από το 2001 δηλαδή και μετά να αναπτυχθεί η απαραίτητη τεχνολογία. Όταν εμείς το 2009 συζητήσαμε τα δικαιώματα των καταναλωτών στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών, είχαμε πει και στο διαβάζω ότι τα κράτη-μέλη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες γεωγραφικού εντοπισμού, οι οποίες θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν προς την υπηρεσία εκείνη η οποία διαχειρίζεται τις κλήσεις εκτάκτου ανάγκης, αμέσως μόλις γίνει η κλήση αυτή και ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλες εκείνες τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Εκτάκτου Ανάγκης 112. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει επιτέλους πού βρισκόμαστε με το ζήτημα αυτό γιατί όσον αφορά τώρα το e-call και τα οχήματα, είναι ένα επιπλέον σύστημα το οποίο θα βασιστεί σε μια υπηρεσία συλλογής πληροφοριών γεωγραφικού εντοπισμού, η οποία κανονικά πρέπει να είναι ήδη διαθέσιμη. Όσον αφορά λοιπόν το επιπλέον κόστος, δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι μεγάλο. Δεν θα υπάρχει ένα μεγάλο επιπλέον κόστος. Το βασικό ζήτημα δεν είναι τόσο η διαθεσιμότητα του δικτύου, αλλά το πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί τα επιπλέον δεδομένα τα οποία θα προέρχονται από τα οχήματα. Και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριο Κόχ πριν από λίγο. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι το ότι θα χρησιμοποιήσει το υφιστάμενο σύστημα καταγραφής ενός ατυχήματος, το οποίο υπάρχει στα οχήματα, που θα είναι εγκαταστημένο στα οχήματα. Στα περισσότερα οχήματα έχετε πλέον ένα πολύπλοκο, αναπτυγμένο σύστημα αερόσακων. Σε ορισμένα οχήματα έχετε 12 διαφορετικούς αερόσακους που δεν ενεργοποιούνται όλοι σε περίπτωση σύγκρουσης. Για παράδειγμα, αν η σύγκρουση είναι μετοπική, θα ενεργοποιηθούν άλλοι αερόσακοι από ότι αν η σύγκρουση είναι στα πλάγια του, οχήματος. Και όπως είπε η κυρία Σεναλόβα, στην ε, παρουσίασή της που είχε κάνει σε ένα σεμινάριο στην Πράγα, φάνηκε τελικά ότι ε, είμαστε σε θέση πολλές φορές να γνωρίζουμε ποια είναι η σοβαρότητα του ατυχήματος. Όλα αυτά τα δεδομένα είναι πολύ σημαντικά και πολύ μπορεί τα δεδομένα αυτά, τα πολύπλοκα και εξειδικευμένα, να δημιουργούν επιπλέον στόχος. Είναι πάντως πολύ σημαντικό να διαβιβάζονται αυτά τα δεδομένα, πιστεύω ότι υπάρχει απαραίτητη τεχνολογία και θα πρέπει οι αρμόδιες εθνικές αρχές να τηρήσουν την συμφωνία την οποία, με την οποία έχουν ήδη δεσμευτεί για την εκμετάλλευση και την διαβίβαση αυτών των δεδομένων. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Δεύτερον, συμφωνώ με την πρόταση που ακούστηκε, ότι το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τους κατασκευαστές των οχημάτων να χρησιμοποιούν το σύστημα επικοινωνιών και για επιπλέον υπηρεσίες υπηρεσίες παροχής περαιτέρω πληροφοριών ή μίσος της λειτουργίας του οχήματος και στις περιπτώσεις όμως αυτές το σύστημα διαβίβαση δεδομένων είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι τα δεδομένα αυτά θα μπορούν να διοχετεύονται παράλληλα χωρίς όμως να παρεμποδίζουν την διαβίβαση των δεδομένων που έχουν να κάνουν με τις κλήσεις εκτάκτου ανάγκη σε περίπτωση ατυχήματος. Νομίζω λοιπόν ότι ε, όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να τα εξετάσουμε. Και από όσο γνωρίζω, Σύμφωνα με τα όσα έχουν αποφασιστεί από τα κράτη-μέλη για τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, οι υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιμες δωρεάν σε όλα τα κράτη-μέλη και σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Φώστερ, ένα από τα πλονεκτήματα του συστήματος είναι ότι σε περίπτωση ατυχήματος είναι απομακρυσμένο μέρος και είναι κανείς μόνος του και ενδεχομένως έχει χάσει και τις αισθήσει του, το σύστημα αυτό θα ενεργοποιήσει αυτόματα την κλίση εκτάκτου ανάγκης που θα επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν το όχημα και τον οδηγό του. Και ενδεχομένω, όπω είπαν και κάποιοι άλλοι ομιλητέ, όπω ο κύριο Μπένιον, θα ήταν καλό να επεκταθεί το σύστημα αυτό. Βέβαια, αν έχει κανεί μαζί του ένα κινητό τηλέφωνο, είτε βρίσκεται σε αγροτικό όχημα, είτε περπατάει, είτε χρησιμοποιεί ποδήλατο, η υπηρεσία γεωγραφικού εντοπισμού ήδη καλύπτεται μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, επομένω θεωρώ ότι δεν θα πρέπει απαραίτητα να εντοπίζεται, να υπάρχει το σύστημα αυτό, να προβλέπεται το σύστημα αυτό στο σύστημα εκτάκτου ανάγκης. Το πρόγραμμα επίσης αυτό το οποίο θα εφαρμοστεί θα πρέπει να είναι απόλυτα συντονισμένο με την τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας, με την τεχνολογία των αυτοκινήτων, καθώς επίσης και με τις υποδομές λήψης των δεδομένων αυτών. Πρέπει να δούμε αν θα καταφέρουμε να συντονίσουμε όλες αυτές τις διαφορετικές τεχνολογίες. Απευθυνόμενος λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να τους ρωτήσω ποιος από από τους τρεις εκπροσώπους των τριών υπηρεσιών θα θέλει να πάρει τον ε, λόγο. Ενδεχομένως ε, η Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας Πληροφορίας θα πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα. Ο κύριος Δαλία λοιπόν έχει πρώτο στο λόγο. Νταβίλα, με συγχωρείτε. Yeah, thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς, οι τρεις υπηρεσίες εδώ Είμαστε σε συνεργασία και αυτό δείχνει πώς η αναγκαιότητα υπάρχει να εργαστούν παράλληλα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αν μου επιτρέπετε, θα μιλήσω και εκ μέρους των άλλων δύο υπηρεσιών της Κομισιόν, της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ επιχειρήσεων, η οποία ασχολείται περισσότερο με το, την υπηρεσία e-call, Εμεί ασχολούμαστε με το θέμα της επικοινωνία και η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ασχολείται με όλη την αλυσίδα και επίσης με το σημείο, με το κέντρο λήψη κλήσεων έκτακτη ανάγκης. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές για την έκθεση και επίσης ε, να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για τις τροπολογίες τους καθώς θα καταστήσουν σαφέστερο το κείμενο. Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν για την Κομισιόν. Εγώ τι θέλω να πω, ότι όπως είπατε κι εσείς, εργαζόμαστε για το ECOL εδώ και πολλά χρόνια και ορισμένες από τις ερωτήσεις που τέθηκαν ήδη έχουν απαντηθεί κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών συνεργασίας, καταρχήν σε επίπεδο έρευνας και κατόπιν ε, μέσω των διαφορών ομάδων και των διαφερόμενων μερών. Τώρα έχουμε και τις ε, πλατφόρμες ECOL, όπου όλοι οι stakeholders συναντώνται και εξετάζουν θέματα που έχουν συζητηθεί, δηλαδή τι θα κάνουμε με τις ε, ψευδείς κλήσεις, πώς θα δημιουργήσουμε ε, ευαισθησία, θα γύρουμε την ευαισθησία κτλ. Σε ό,τι αφορά το θέμα της τυποποίησης και τη τεχνολογική σκοπιά, είναι έτοιμη να αναπτυχθεί η υπηρεσία, αλλά φυσικά όπως υπόθηκε εδώ, υπάρχει και η ανάγκη και τα τρία τμήματα να συνεργαστούν για να έχουμε ταυτόχρονη εφαρμογή και αυτό κάνουν οι υπηρεσίε της Κομισιόν. Τώρα, θέσατε δύο συγκεκριμένα ζητήματα σε σχέση με την ε, κατάσταση με το στάτους ε, ε, της τοποθεσίας αυτό ανήκε στην ε, ε, οδηγία της καθολικής υπηρεσίας. Ε, τώρα με την νέα τροπολογία του 2009 έχουμε επαναλάβει και ενισχύσει αυτή την υποχρεωσία. Έτσι λοιπόν η κατάσταση εξαρτάται από τη μία χώρα στην άλλη και έχουμε ορισμένες χώρες όπου τη στιγμή της έλευσης της κλήσης 112 ε, κάποιοι πάροχοι μπορούν να δουν την τοποθεσία στην οθόνη, δηλαδή υπάρχει ε, ε εντοπισμό, ταυτοποίηση από το, του κινητού. Αν μιλήσουμε τώρα για τις απομακρυσμένες περιοχές, ε, τότε το e-call ε, θα βασίζεται, ε, θα έχει μεγαλύτερη ακρίβεια γιατί θα βασίζεται σε εντοπισμό τοποθεσία μέσω δορυφόρου. βέβαια, σε αγροτικές περιοχές θα έχουμε διαφορετικό επίπεδο ακρίβειας. Σε ορισμένα κράτη-μέλη ήδη έχει ε, υλοποιηθεί αυτό, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετική προσέγγιση και δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει αυτή τη δυνατότητα του core location. Και το διερευνούν αυτό κάποιοι συνάδελφοι. Υπήρχε και το ερώτημα, ζητήθηκε από την Κομισιόν να δώσει μεγαλύτερο input από τις μελέτες. Έχουμε τη μελέτη αντικτύπου, όπου εξετάσαμε όχι μόνο τα δεδομένα, αλλά εξετάσαμε και άλλες μελέτες που έχουν ήδη γίνει. Καλύπτεται όλο το κόστος ε, και για το, τηλεπικοινωνία και για την υποδομή και για το όχημα και υπολογίσαμε το πιθανό κόστος και τα ωφέλη και το αποτέλεσμα είναι για την υποχρεωτική εισαγωγή του e-call ε, η αναλογία κόστος ωφέλους θα είναι κάτι είναι θετική. Για τα υπόλοιπα δύο, ε, ο εκούσια προσέγγιση είναι να το αφήσουμε στην αγορά δεν ε, ίσχυε κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν ε, αρχίσαμε να βλέπουμε τον αντίκτυπο στο κόστος του οχήματο ανάλογα με τα διάφορα είδη ατυχήματο. Ήρθαμε σε επαφή και με διάφορα διαφορούμενα μέρη, με τους ε, κατασκευαστές και προσπαθούμε επίσης και σε επίπεδο προτύπων να εντοπίσουμε ποια θα μπορούσε να είναι η ελάχιστη λύση που θα μπορούσε να παρουσιάσει το ελάχιστο σετ δεδομένων στα κέντρα έκτακτης ανάγκης και επίσης θα μπορούσε να έχει και όσο το δυνατόν λιγότερο αντίκτυπο στην ε, αλυσίδα των αξιών. Και έτσι λοιπόν καταλήξαμε στο πρότυπο που έχουμε παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Και αυτά τα έγγραφα είναι διαθέσιμα, νομίζω ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση και συνάδελφοι. Αν έχετε τα δεδομένα, η κυρία Φώστερ αναφέρθηκε στο κόστος ε, για το όχημα. Μήπως μπορείτε να μας ε, πείτε ποια υπόθεση κάνετε σε σχέση με την εγκατάσταση του εξοπλισμού στα αυτοκίνητα, στη μελέτη δικτύπου σας. Βεβαίω. Καταρχήν, ε, το να κάνει κανείς μια υπόθεση για το κόστος είναι κάτι δύσκολο, γιατί έχουμε όλο το περιβάλλον τη αγορά και ενίοτε οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν είναι έτοιμες να μας δώσουν αυτά τα νούμερα. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει τεχνολογία και έχει εφαρμοστεί ήδη σε ιδιωτικά οχήματα, αλλά μέσω και του πολιτικού προγράμματος είδαμε ότι ε, χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένες χώρες και έτσι λοιπόν ορισμένες χώρες μπορούν να λάβουν αυτό το e και να το διαχειριστούν. Τώρα μιλήσαμε με του διάφορου προμηθευτέ. Ε, λόγω τη οικονομία κλίμακα θα μπορούσε να, το κόστο να φτάνει στα 50-60 ευρώ. Για τη μελέτη δικτύπου εξετάσαμε και το διάφορα είδη κόστου ε, που σχετίζονται με την έρευνα, με το σχεδιασμό και την ενσωμάτωση. Και επίσης έχουμε και τον παράγοντα πολλαπλασιασμού επί τρία. Έτσι λοιπόν για τη μελέτη αντικτύπου, λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την αρχική υπόθεση ότι η συσκευή θα κοστίζει 50-60 ευρώ επιπλέον, έτσι λοιπόν το πρόσθετο κόστος ε, για το όχημα θα ήταν περίπου 180 ευρώ. Αυτό εξετάσαμε στη μελέτη δικτύπου. Αυτό το κόστος δεν είναι προαιρετικό. Ε, στην ε, περίπτωση που έχουμε ε, υποχρεωτική εισαγωγή, αυτό θα είναι διαφανές ε, για τους χρήστες Όπω, ε, παραδείγματο χάρη τώρα με τι ζώνες ασφαλεία. Κανεί δεν ξέρει πόσο πληρώνει επιπλέον για να έχει το όχημα ζώνη ασφαλεία. Ε, και έτσι λοιπόν ε, το ίδιο θα συνισχύει και για με τη συσκευή του e-call. Κύριε θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Από την γάμα Move θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Όχι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ να επανέλθω είτε στους ευρωβουλευτές είτε στους συζητητές αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση. Κύριε Φώστερ. Δεν θέλω να είμαι αγενής κύριε Πρόεδρε, αλλά η Επιτροπή αντιλαμβάνομαι ότι ε, θα μας ε, απαντήσουν όταν θα τεθεί το ερώτημα. Δηλαδή ο πολιτικός πρέπει όλα αυτά να τα συζητήσει διεξοδικά με την εμπλεκόμενη βιομηχανία και καταλήγουμε ε, στο πώς πρέπει να εισαχθεί μία βιομηχανία. Αλλά η βιομηχανία μπορεί να καταλήξει σε ένα τελείως διαφορετικό αριθμό. Δεν ξέρω ποιον οι αριθμοί είναι σωστοί διότι εγώ έχω μιλήσει σε πολλές εταιρείες εταιρείε ε, σε βάθος χρόνου και βλέπω, όπως είπα και πολύ σαφώς στις παρατηρήσεις μου, ότι προφανώς όσο περισσότερα μηχανήματα παράγεται, τόσο θα πέφτει η τιμή. Αλλά μιλάμε στην αρχή για 300 ευρώ ή 300 λίρες για να ξεκινήσουμε. Δεν είναι 30 ευρώ ή 50 ευρώ, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένα κόστος και για τη βιομηχανία ε, μπορείτε βέβαια να πείτε ότι θα το χάσουν ε, από την τιμή του αυτοκινήτου αλλά όλα τώρα πολλούνται διεθνώς και κάθε κόστος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη γενικότερα δεν μιλάμε για πενταροδεκάρες και ε, ε, πρόκειται για μία βιομηχανία πολύ σημαντική και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Δεν θέλω να ανοίξω μια συζήτηση, γιατί αυτό που είναι βασικό είναι να μας στείλετε τα στοιχεία σας και έχω τα στοιχεία της βιομηχανίας που εμπλέκεται μπροστά μου. Απλώς θα ήθελα να σας πω ότι όταν μιλάω για το κόστος και τα στοιχεία που μας έδωσε η αυτοκινητοβιομηχανία σας είπα ότι δεν είναι εύκολο να έχουμε ακριβή στοιχεία για τους διάφορους παίκτες αλλά από το, την αυτοκινητοβιομηχανία έχουμε λάβει στοιχεία και λέμε στην ε, μελέτη επιπτώσεων δεδομένων ποια είναι τα στοιχεία που μας έχουν δώσει οι προμηθευτές ε, και ε, πολλές φορές η αυτοκινητοβιομηχανία αυξάνει τις τιμές όταν μιλά για την εισαγωγή ενός τέτοιου συστήματος Οπότε εξετάσαμε τις προσφορές των διαφόρων προμηθευτών και θα δείτε στην μελέτη επιπτώσεων ένα κεφάλαιο που αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το θέμα. Νομίζω το καλύτερο είναι να μας ξαναστείλετε τις ε, προϋποθέσεις σας και θα τις διαβάσουμε με μεγάλη προσοχή. Τώρα λοιπόν παρακαλώ τους δύο εισηγητές να λάβουν τον λόγο και να συνοψίσουν και να ε, επιβεβαιώσουν ότι θα συνοψιστούν οι τροπολογίες για την ε, για την ψηφοφορία στην την 3η 19 Ιουνίου αυτή είναι η ημερομηνία που ξέρω και θα πρέπει να έχουμε λήξει ε, να έχουμε επεξεργαστεί τροποδογίες πλήν η κυρία Σανίλοβα έχει καταρχήν το λόγο Σας ευχαριστώ πρόεδρε θα είμαι πολύ σύντομη Καταρχάς, να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης ηγητές και όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, πληροφορίες και τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις θετικές αλλά και αρνητικές σας παρατηρήσεις και για τις τροπολογίες βέβαια που έχετε καταθέσει. Ξέρω ότι η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και ότι καλύπτει πολλές τεχνικές πτυχές. Προσβλέπω ουσιαστικά σε μια θετική συνεργασία, καθώς επίσης και σε περισσότερες τροπολογίες και σε, στην έβρεση συμβαστικών τροπολογιών. Ο κύριος Κόχα. Και εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση. Πιστεύω ότι τα περισσότερα συνοψίζονται σε τρία συστήματα. Διαθεσιμότητα, ε, ε, ε, κίνηση της κλίσεως και ανταπόκριση. Όπως η αερόσακη. Υπάρχουν βασικά θέματα τα οποία θα συμβούν στο αυτοκίνητα και ε, γι' αυτό πρέπει κανείς ε, να ε, αξιολογήσει θετικά την έκθεση, να διώξει τις, τις χρήσεις οι οποίες δεν ενδείχνονται και βάσει του χρονοδιαγράμματος θα προχωρήσουμε και θα τα επεξεργαστούμε. Ευχαριστώ όλους αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν και την ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσβλέπουμε στο να συναντηθούμε για να ε, συζητήσουμε την πρότασή σας και αυτή τη βασική έκθεση. Είναι μία έκθεση κατά πρωτοβουλία, πρόκειται για πολιτική έκθεση και θα δούμε τι θα αποφασίσει να κάνει η Επιτροπή και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει και σε συζήτηση με τα κράτη-μέλη διότι πολλά έχουν συζητηθεί. Ευχαριστώ και λίγη κοινή συνεδρίαση. Η Επιτροπή της κοινή Αγοράς θα επανέλθει στις 3 το απόγευμα για, καταρχήν με τις δημόσιες προμήθειες και λύεται η συνεδρίαση.